Yeah. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, <clears throat> να συνεχίσουμε την απογευματινή συνεδρίαση με λογική απόψεων σε σχέση με την ε, πορεία των εμπορικών σχέσεων της Νορβηγίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας παρακολουθήσω να κάνετε λίγο ησυχία. Από τη δική μου σκοπιά πρέπει να επικεντρωθούμε στα πρόσφατα μέτρα της νορβηγικής ε, κυβέρνησης ε, φαίνεται ε, να είναι προστατευτικά και αναφέρομαι ε, στο, στο 72% ε, δασμούς εισαγωγικούς που έχουν βάλει σε ορισμένα είδη κρέατος και τυριού και στο προσχέδιο προπολογισμού του 2013 η νορβηγική κυβέρνηση πρότεινε από ειδικού δασμούς να περάσουμε σε ad δασμούς για κρέας και προϊόντα τυριού και σύμφωνα με την Επιτροπή, με τη ΓΑΜΑ Άγκρη, ε, θα φυγούν τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περισσότερες φορές το πρόβιο κρέας. Ε, ο προϋπολογισμός ε, στην... πρόκειται να σήμερα από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο έτσι λοιπόν καλέσαμε τον ε, κύριο Λέικφολ, ε, τον πρέσβη της Νορβηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ να το, το καλωσορίζουμε ένθερμα στην Επιτροπή μας. Σας καλέσαμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε την νορβηγική προοπτική και να ανταλλάξετε απόψεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο, καταρχήν εσείς κύριε Πρεσβευτά, και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και την ευκαιρία να απευθυνθώ σε αυτή την Επιτροπή. Με την ε, ανοχή σας ε, θα σας απασχολήσω λίγα λεπτά για τρία σημεία. Το ένα θα είναι η ευρεία προοπτική στις συνολικές σχέσεις μας γενικά. Δεύτερο σημείο θα αναφέρεται στη Γεωργία και το τρίτο σημείο θα αναφέρεται στα θέματα που αναφερθήκατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Καταρχήν, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας δώσω ορισμένα κυρία στοιχεία. Η Νορβηγία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νορβηγία τα τεταρτά του αλλά το εμπορίου μας ε, ε, είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενέργεια 20% των συνολικών αερίων, του συνολικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από την Νορβηγία και το πετρέλαιο 12%. Αναφέρω αυτά τα τεχνητικά στοιχεία για να σας δείξω το μέγεθος ε, των οικονομικών μας σχέσεων και τη σημασία που έχουν προφανώς για την Νορβηγία, αλλά ήθελα να πω και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη με ορισμένες εξαιρέσεις στις ε, σχέσεις μας ε, διέπονται από την ε, Συμφωνία ΕΟΧ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που επιτρέπει στην Νορβηγία να συμμετέχει πλήρως στην εσωτερική αγορά, κάτι που ισχύει από το 1994. Φυσικά, όντας μέρος ε, της ε, ενιαία αγοράς, ε, ξεπερνά την οικονομία, αφορά τους ισότιμου κανόνες για τις επιχειρήσεις, για τα άτομα, για τους εργαζομένους, για του φοιτητέ. Και χθε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΕΟΧ, όταν κάναμε μια κοινή αξιολόγηση για το πώς λειτουργήσε είπε το Συμβουλίο και παραθέτω ε, ενώψη της 20ης επαιτίου της ε, νέας αγοράς ε, στο τέλη του φετινού χρόνου το Συμβουλίο αναγνωρίζει με ικανοποίηση ότι η Συμφωνία ΕΟΧ ήταν ε, ένα καλό μέσο για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό συμπίπτει πλήρως ε, με την αξιολόγηση της νορβηγικής κυβέρνησης στη Λευκή Βιβλίου που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα στο Κοινοβούλιο πιστεύουμε με τη συμφωνία εξυπηρέτησε καλά όλα τα μέρη και η κυβέρνηση δηλώνει ότι αυτή είναι η φιλοδοξία της Νορβηγίας στο μέλλον να συνεχίσει να αναπτύσσει μια δυναμική σχέση σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, συνολικά, και δεν ολοκληρώνω το πρώτο μου σημείο, νομίζω ότι είναι ορθό να πούμε ότι οι σχέσει μεταξύ Νορβηγία και Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικά και πολιτικά, είναι πράγματι καθολικέ και δυναμικέ. Και μα έχουν εξυπηρετήσει καλά αυτέ οι σχέσει. Τώρα, να περάσω στη Γεωργία. Αναφέρθηκα στην φράση με κάποιε εξαιρέσει ο ΕΟΓΔΙΕΠΗ τη σχέση μα. Η Γεωργία είναι μια τέτοια εξαίρεση. Οι διατάξεις της συμφωνίας δεν περιλαμβάνουν τη Γεωργία. Η Γεωργία χρειάζεται ένα καθεστώς ε, ε, input που να επιτρέπει μια ε, βιώσιμη εγχώρια παραγωγή. Δεν είμαστε μόνοι στην κατηγορία αυτή. Νομίζω ότι οι περισσότερες χώρες ανήκουν εκεί. Το δικό μας καθεστώς αντικατοπτρίζει το σημείο φετηρίας μας, όπως θα το έλεγα, για την αγροτική παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, Προφανώς ε, συμμετείχαμε σε διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, και μπήκαμε σε εμπορικές διευθετήσεις και στον ΠΟΕ και στο πλαίσιο του ε, ΕΟΧ αναφέρομαι στο άρθρο 8 πρωτοκόλλο 3 και στο άρθρο 19 το άρθρο 8, σύμφωνα με το άρθρο 8, η Γεωργία δεν διέπεται από τις Γενικές Συμφωνίες και το πρωτόκολλο 3 διέπει το αμοιβαίο εμπορίο μα στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και το άρθρο 19 μας υποχρεώνει να πετύχουμε προοδευτική απελευθέρωση στα γεωργικά προϊόντα, στον πορείο γεωργικών προϊόντων. Όμω. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες συνθήκες για να γίνει αυτό. Θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο των αντίστοιχων γεωργικών πολιτικών και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα ε, και θα πρέπει να γίνει σε μια αμοιβαία διμερή βάση που να ωφελεί και τους δύο. Πιστεύω ότι η Νορβηγία ε, έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές. Μπήκαμε σε επιτυχείς κύκλους ε, αναθεωρήσεων και διαπραγματεύσεων που επέτρεψαν σημαντικές επαναχωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο γύρος παραχωρήσεων εφαρμόστηκε την 1η Ιανουαρίου 2012 και περιλάμβανε μεγάλες ε, παραχωρήσεις όπως ε, τη της ποσόστοσης ε, για το τυρί. Αν δείτε ε, τις εξαγωγές από την Ορβηγία, <clears throat> σε αγρογεωργικά προϊόντα έχει αυξηθεί οι εισαγωγέ μα, μα συγχωρείτε, έχουν αυξηθεί 100% ενώ οι εισαγωγέ μα 45%. Δεν είναι κλειστή η αγορά τη Νορβηγία. Το 50% τη συνολική μα κατανάλωση προέρχεται τι εισαγωγέ και από αυτέ τι εισαγωγέ το 70% προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε να πείτε λοιπόν ότι πάνω από το 1 τρίτο της συνολικής μας κατανάλωσης ε, στην Νορβηγία προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε κάτι που είπε ένας ε, δανός ε, φιλόσοφος, αλλά όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη μεγέθυνση αυτή της αγοράς ε, για να ωφεληθούν η εγχωρή παραγωγή αλλά και η εξαγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Και τέλος, συγκεκριμένα η αναφορά στα σημεία που θίξατε εσείς εισαγωγικά. Θα ήθελα να κάνω μια σαφή διάκριση μεταξύ το ε, το, για το θέμα της αλλαγής ε, από συγκεκριμένους δεσμούς ε, με το, σε άλλους δεσμούς με το δυναμικό. Τώρα, εδώ δεν είχαμε αλλαγή του δεσμού, αλλά είχαμε αλλαγή της κατηγοριοποίησης δεσμολογικής κατηγοριοποίησης για αρκετό καιρό είχαμε λάθος εφαρμογή σε αυτό το τομέα. Δεν είμαι τεχνικός εμπειρογνώμονας, αλλά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για με μακροφύλλα για πολλά καιρό, ε, όλη τη δεκαετία του 90, εισαγάγαμε ε, αυτό το φυτό ως λουλούδι και εν μέρει ως θάμνο που είναι αδεσμολόγητο. Και για πολλά χρόνια οι εισαγωγέ του φυτού θεωρούνταν ως θάμνος, ενώ οι νορβηγικές τελωνιακές αρχές το συνειδητοποίησαν, έλαβαν μία διοικητική απόφαση, έτσι ώστε η κατηγοριοποίηση, η ταξινόμηση ε, να επανέλθει σε αυτό που έπρεπε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να αναγνωρίσω ότι οι εξαγωγείς οι οποίοι μπορούσαν να λανθασμένα ε, να εξάγουν με μηδέν δασμό, αδασμολόγητα ε, ήταν ικανοποιημένοι όταν ε, υπήρξε αυτή η τροποποίηση. Αλλά αυτή ήταν μια διοικητική απόφαση, δεν είχε καμία σχέση με πολιτικές αποφάσεις από την Ορβηγική κυβέρνηση. Η αλλαγή από τον ειδικό δασμό σε advalorem. Στον προϋπολογισμό του 2013 η κυβέρνηση πρότεινε έξι δασμολογικές γραμμές για τη ρή, πρόβιο κρέα και βίο να αλλάξουν από ένα συγκεκριμένο δασμολογικό ποσοστό σε advalorem δασμό από την 1η Ιανουαρίου 2013. Δεν ξέρω αν η απόφαση αυτή ελήφθη, αλλά όπως σωστά αναφερθήκατε και εσείς στην εισαγωγή σας, το Κοινοβούλιο θα λάβει μια απόφαση για το συνολικό προϋπολογισμό σήμερα. αυτή η αλλαγή συνάδει πλήρω ε, με τις υποχρεώσεις μας στον ΠΟΕ κατόπιν του κύκλου της Ρουάη. Μπορούσαμε να επιλέξουμε αν θα έχουμε ειδικού δασμούς ή αν θα έχουμε αντιβαλόρεμ. Τότε είχαμε αποφασίσει να έχουμε ειδικού δασμούς. Με το πέρασμα των χρόνων, ε, το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτών των ειδικών δασμών διαβρώθηκε. Και αυτό είναι το ιστορικό της πρότασης ε, που έθεσε η κυβέρνηση του Κοινοβουλίου. Οι αλλαγές προτείνονται με έναν τρόπο που να ελεγχιστοποιούν ε, τις αρνητικές συνέπειες ε, και να μην απειλούν σημαντικά τις παραχωρήσεις που παραχώρησε η Νορβηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανωμένου και συμπεριλαμβανομένων και των 7.249 τόνων αδεσμολόγητων για το τυρί και 900 τόνων για το κρέας. Οι δικοί μας ε, υποχρεώσει απορρέουν από το άρθρο 19 και δηλώνουν ότι η προοδευτική απελευθέρωση του γεωργικού εμπορίου θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των αντίστοιχων γεωργικών πολιτικών των μερών και σε μια αμοιβαία βάση. Εμείς συνεχίζουμε να ακολουθούμε τις προθέσεις ε, του άρθρου 19 και αυτό μας επέτρεψε την αύξηση 150% εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Νορβηγία από το 2000. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τις διαδικασίες που αναφέρονται στη Συμφωνία ΕΟΧ. Χθες, όπως είπα, είχαμε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου ΕΟΧ και στα συμπεράσματα, στα κοινά συμπεράσματα της συνεδρίασης αυτής, Λέγεται ότι το Συμβούλιο ΕΟΧ ε, αναμένει την επόμενη αναθεώρηση το 2013-2014 των ε, κριτηρίων που θα διέπουν το είναι εμπορία γεωργικών προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Νορβηγία, προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει στα πλαίσια του άρθρου 19. Αυτά είχα να πω εγώ, Πρόεδρε. Προσπάθησα να είμαι σύντομο και να σας παρουσιάσω μια ευρεία εικόνα και το ιστορικό της γεωργικής πολιτικής και προσπάθησα να σας παρουσιάσω τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε, Πρέσβη, για αυτή την επισκόπηση. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Λίκ Ντομαρτή που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη, τον κύριο Λίκ Ντεβίνιε που εκπροσωπεί την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συγχωρείς, Λίκ. Όμως θα σε παρακαλούσα να μας δώσεις και τις δικές σου απόψεις για το όλο θέμα. Και επειδή ο πρέσβης έθιξε το ζήτημα των ελεύθερων ποσοστώσεων, σε παρακαλώ να μας εξηγήσεις το, το σύστημα των ε, δασμών για τις ελεύθερες ποσοστώσεις. Όσοι κάνουν εξαγωγές βάσει αυτών των ποσοστώσεων θα πάρουν κάτι, θα πρέπει να πληρώσουν κάτι. Πώς γίνεται ακριβώς, ποια είναι η ερμηνεία σου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη διαφήμιση. Βεβαίως δεν διαφωνούμε με τον πρέσβη γιατί και εμείς λέμε ότι έχουμε καλές και σταθερές και ε, υγιείς σχέσεις με την Ορβηγία, τον πέμπτο κατά σειρά εμπορικό μας εταίρο. Βεβαίως, καλύτερα να βλέπουμε προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν εκ των προτέρων παρά να ενσκύπτουμε στα προβλήματα. Γι' αυτό εφόσον έχουμε 36%, 36 δισεκατομμύρια έλλειμμα σε σχέση με τι εμπορικέ μας σχέσεις με την Ορβηγία, σίγουρα οι σχέσει αυτέ είναι πιο υποφελείς για την ίδια τη χώρα. Πάντως, χθε στις συζητήσει του Συμβουλίου που ασχολούνται με το θέμα αυτό, τα θέματα αυτά συζητήθηκαν και δεν συμφωνώ με τον πρέσβη ότι τα μέτρα αυτά είναι ή προστατευτικά ή ότι σκοπός δεν ήταν να είναι προστατευτικά και εάν αυξηθεί ο δασμός από 0 σε 72% είτε το αποκαλέσει κανείς διοικητικό μέτρο, τελωνιακή απόφαση, ε, διοικητική απόφαση είναι μέτρο προστατευτισμού. Και τελικά θύματα θα είναι η καημένοι η Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι νορβηγοί τελωνιακοί να ξεχωρίσουν το τύπο 1 από το τύπο Α από το τύπο Β. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια έκαναν ένα τέτοιο λάθος. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα δασμό του 72%. Όσο για τα άλλα προϊόντα που συζητήθηκαν, το τυρί, η αύξηση είναι δεκα, δεκαπλάσια για το ε, κρέας πενταπλάσια η αύξηση και για τα αυγά διπλάσια και αυτό μας ε, δυσαρεστεί ιδιαίτερος ιδίως για το τυρί δεν νομίζω ότι είναι καταλληλότερη χρονική στιγμή να δυσκολέψουμε κι άλλο την ζωή των εξαγωγών μας. Βεβαίως, η Νορβηγία αποφελείται πλήρως από τις εμπορικέ σχέσεις με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ε, θίξει τα θέματα αυτά με πολλές σε πολλές συναντήσεις με τους νορβηγικούς εταίρους. Ε, τον Νοέμβριο ο Επίτροπος Όλος συνάντησε τον Υπουργό Γεωργίας, τον ομολογό του. Ε, Χθε υπήρξε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Νορβηγία και εκφράστηκαν οι βαθιέ μα ανησυχίε και η ε, λύπη μα για την ε, κακή επιλογή, τη χρονική επιλογή για την ενίσχυση του προστατευτισμού. Και το Συμβούλιο, χθε τα συμπεράσματά του, εξέφρασε τι απόψει του κατά τη ενίσχυση του προστατευτισμού. Τα νορβηγικά μέτρα λοιπόν είναι πραγματικά τελείω κακοδεχούμενα αυτή τη στιγμή. Ο πρέσβης παρέθεσε και μια πρόταση των ε, ε, συμπερασμάτων του Συμβουλίου χθες. Αλλά η επόμενη φράση που ξέχασε λέει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λυπάται για την πρόταση της νορβηγική κυβέρνησης να αυξηθούν οι τελωνιακοί δασμοί περνώντας από, του από τους συγκεκριμένους ειδικού δασμούς σε ειδικού δασμούς ε, επί γεωργικών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την ε, Νορβηγία και την παροτρύνει να αναστρέψει την απόφαση αυτή. Είναι μια ολόκληρη παράγραφος και το, το απόσπασμα από το οποίο μας ανέφερε ο πρέσβης. Κάποια λεγόμενα. Για να μην αντιφάσκουμε λοιπόν με το πνεύμα της συμφωνίας, πρέπει να πούμε ότι και η μορφή της ε, διάταξης μας βρίσκει αντίθετος. Το άρθρο 19 είναι σαφές. Τα μέρη της συμφωνίας θα πρέπει να εξετάσουν κάθε ανομαλία που θα προκύψει στις σχέσεις ως προς τα γεωργικά προϊόντα. Και δεν νομίζουμε ότι όταν μονομερός έλαβαν μέτρα η Νορβηγία εταιρεία κάτι τέτοιο. Ε, επίσης, τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ε, πετύχουν την πλήρη εξομάλυνση του γεωργικού εμπορίου. Δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε σε κανέναν τι να κάνει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε επίση ότι η αύξηση του δασμού από το 0 στο 72% ή δεκαπλασιασμό ή ο διπλασιασμό ή ο τριπλασιασμό δείχνει ότι θα φτάσουμε σε συνολική εξομάλυνση του γεωργικού εμπορίου. Βάσει τη συμφωνία αυτή πάλι έχουμε υποχρέωση να συναντώμαστε αναδυνατία και έχουμε συναντηθεί μόλον δύο φορέ από το 1993 για να συζητήσουμε για τα προϊόντα αυτά. Ολοκληρώνοντα λοιπόν, θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά αντίκεινται και στο πνεύμα και στην μορφή, το περιεχόμενο ακριβώ, το σώμα τη συμφωνία. Ζητούμε από την Ορβηγική κυβέρνηση να στείλει τη συμφωνία, τα μέτρα που μονομερό αποφάσισε. Και βεβαίω αφήνουμε τη δυνατότητα νομικής προσφυγής ανοιχτή. Επίσης, Πρόεδρε, για να απαντήσω και στις δικές σας ε, απευθείας ερωτήσεις, αυτή τη στιγμή το σύστημα των ποσοστώσεων το, διαχειρίζεται ένας, ε, το διαχειριζόμαστε βάσει μηχανισμού διαγωνισμών. Ο πρώτος διαγωνισμός για το 2011 για το τυρί οδήγησε σε δασμό 24,98 νορβηγικών κορονών ανά κιλό. βάση και του βασικού δασμού για το πλέον προτιμόμενο έθνος του νορβηγικού συστήματος. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της, την ηχόπη των συνέβησαν στο Συμβούλιο, ο κύριος Χέλνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που <clears throat> ήρθε κοντά μας ο ε, πρόεδρος της Νορβηγίας με την πολυάριθμη αντιπροσωπεία του. Έχουμε στενές ε, εμπορικές σχέσεις, έχουμε συνάψει πολλές συμφωνίες και σε αυτή την Επιτροπή ε, δεν έχουμε μιλήσει αρκετά για τη σχέση με την Νορβηγία. Γι' αυτό λοιπόν είναι λυπηρό το γεγονός ότι η αφορμή της σημερινής επίσκεψης ε, είναι ε, το πρόβλημα που υπάρχει με τους ε, δασμούς στην Νορβηγία, οι οποίοι επιβλήθηκαν χωρίς να έρθουν οι Νορβηγοί ε, σε επαφή 290, στο τυρί, ε, στο 344 στο κρέας και 494% υπάρχουν και αυτοί οι δεσμοί πραγματικά υπέρογκα ποσά. Ε, στην πράξη λοιπόν σημαίνει το εξής. Μίλησα με Σουηδούς γαλακτοπαραγωγούς. Κατ' ουσίαν οι Σουηδοί δεν μπορούν πλέον να εξάγουν τυρί από τη Σουηδία προς τη Νορβηγία. Διότι ε, το είδατε και χτες αυτό, ήταν εδώ η γαλακτοπαραγωγή και η Νορβηγή και αυτοί πρόκειται να αντιμετωπίσουν ε, προκλήσεις. Δεν είναι όμως ε, οι μόνοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν είναι δικό τους το πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο αυτοί το πρόβλημα στη Γεωργία. Ίσως θα μπορούσε ε, να υπάρξει ε, κατάργηση του προστατευτισμού χωρίς ε, να καταργηθεί και το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νορβηγία. Διάβησα στον Economist, υπάρχει και ένα άρθρο για την νορβηγική οικονομία, πάρα πολύ ωραία, αυτά που αναφέρονται. Περίπου 5% είναι η ανάπτυξη στη χώρα, αυτό στις Βρυξέλλες τα ακούμε σχεδόν ποτέ, σπάνια έως ποτέ. Ε, η ανεργία ε, είναι επίσης ε, πάρα πολύ χαμηλή, περίπου στο 3%, άρα δηλαδή υπάρχει εμπορικό πλεόνασμα. Κατά κανόνα λοιπόν τι συμβαίνει. Ο προστατευτισμός προκύπτει μετά από οικονομική κρίση. Αλλά σας ερωτώ, στην Ορβηγία Πού είναι η κρίση σας, γιατί λοιπόν εισάγετε μέτρα προστατευτισμού ή μήπως αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κάνετε όλα αυτά ε, στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας, ότι οι στόχοι είναι πολιτικη ε, πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, έχουμε το άρθρο 19.2 που αναφέρει ότι οι συμβαλόμενοι θα καλούνται μακροπρόθεσμα να επιφέρουν ε, σταδιακή απελευθέρωση στο οικονομικό εμπόριο. Αυτό είναι ο στόχος. Και γι' αυτό λοιπόν διαρωτώ με κι εγώ με ποιο τρόπο συμβάλλετε εσείς ε, στην ε, απελευθέρωση των γεωργικών προϊόντων. Αυτά τα οποία μας είπε ο πρέσβης είναι ενδιαφέροντα. Χρησιμοποιείς τη λέξη αμοιβαιότητα πάρα πολύ ωραία, αλλά τι σημαίνει η αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα δηλαδή να εισάγουμε κι εμείς δασμούς και προς αμοιβαίο όφελος, είπατε και αυτό. Τώρα, ποιο είναι το αμοιβαίο όφελος σε αυτά τα οποία κάνατε. Ίσως ε, αυτά τα οποία λέω να έχουν ε, λιγάκι προσωπική, σαν προσωπική επίθεση, αλλά Ξέρετε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πω ότι θα ήταν καλό να είστε και εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιφέρετε την δική σας την ε, τεχνογνωσία. Εγώ ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Εμπορίου, πάντα υπερασπιζόμουν τις ε, νορβηγικές επιχειρήσεις και είχαμε και μία αντιπαράθεση με την Κομισιόν για τον Σολομό της Νορβηγίας, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε την υπόθεση. Εγώ λοιπόν έχω περασπιστεί επανειλημμένα την Νορβηγία και γι' αυτό νιώθω μεγάλη απογοήτευση για το ότι η Νορβηγία εισάγει προστατευτικά μέτρα χωρίς να μπορεί να εξηγήσει γιατί. Αυτά δεν είναι τεχνικής φύσεως ε, θέματα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Γιατί λοιπόν στο μέλλον εγώ να ξαναυπερασπιστώ την Νορβηγία. Εάν λοιπόν η Νορβηγία δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα στους γαλακτοπαραγωγούς, ε, και εγώ δεν θα την ξαναπερασπιστώ. Ευχαριστώ. Κριστοφέρ, αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, να κάνω κι εγώ κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις. Δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Κοιτάξτε, αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα στο θέμα αυτό είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ενδεχομένως να μπορεί να σταθεί νομικά, όπου βέβαια και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν εξέφρασε τις εμβολίες του, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι το τι είναι νομικά εφικτό και το τι είναι, τι ήθιστε να συμβαίνει ανάμεσα σε φίλους την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους θα, θα τεθεί κάτι σε ισχύ στη Νορβηγία, ε, το οποίο όχι μόνο είναι παράνομο, αλλά είναι και ασυνήθιστο ανάμεσα σε φίλους. Εμείς ε, θα προτιμούσαμε να συζητήσουμε προηγουμένως και δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Όλοι λοιπόν όσοι ασχολούνται με γεωργικά προϊόντα γνωρίζουν πολύ καλά ότι ειδικά στον τομέα της γεωργίας υπάρχουν ευαίσθητα προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνω λιγάκι αυτά ε, που συμβαίνουν στον τομέα του κρέατος. Αλλά δεν νομίζω ότι ε, τα γαλακτοκομικά και τα τυριά είναι ευαίσθητο προϊόν. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα προτιμούσα να είστε λιγάκι πιο προσεκτικοί. Και αυτό που επίσης κατέστησα φες, κύριε Πρέσβη είναι οι αδασμολόγητες ποσοστώσεις αλλά στην πραγματικότητα οι ποσοστώσεις αυτές δεν είναι αδασμολόγητες. Αυτό που είναι αδασμολόγητο, το είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ε, είναι αντικείμενο δημοπρασίας ε, στην αγορά. Και μετά οι τιμές ε, προσαρμόζονται ανάλογα με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Δεν ξέρω πουθενά στον κόσμο να μην ισχύει αυτό το σύστημα των ποσοστώσεων. Δηλαδή και τα, δασμολόγητα ε, προϊόντα κατ' ουσίαν ε, τελικά δασμολογούνται. Είναι πολύ κανονιστικό αυτό που κάνετε. Είναι σαφώς ε, μέτρο προστατευτισμού. Και αυτό δεν το θέλουμε, το έχουμε συμφωνήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ήμουν ευγνώμων εάν λαμβάνατε υπόψη σας την άποψη της Επιτροπής που έχουν γίνει ήδη κάποιες συζητήσεις αλλά και των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου ε, που εκφράστηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως δεν πρόκειται για επίσημη θέση του Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω ότι συνειδητοποίησατε ότι ε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Ο κύριος Σόλτς παρακαλώ έχει το λόγο. Κοιτάξτε, θέλω να κάνω και εγώ μια παρατήρηση, η οποία θα έπρεπε λιγάκι να μας ε, προβληματίσει. Πριν από αρκετό καιρό, εδώ στην Επιτροπή μας, μιλήσαμε για τις ε, διαπραγματεύσεις, είχαμε μια σχετική έκθεση, ψηφίσαμε από αυτή και τέθησαν κάποιες, ε, το θέμα κάποιων εξαιρέσεων. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, το όλο θέμα είναι το εξής. Δεν υπάρχουν ακριβή οι διαπραγματεύσει δεν είναι ακριβεί. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η άλλη πλευρά θα πρέπει με απόλυτη διαφάνεια να ορίζουν το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, τι επιτεύχθηκε, που υπάρχουν προβλήματα, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να δούμε τι γίνεται ε, όταν υπάρχουν εξαιρέσεις. Εντάξει, θα τις δεχόμαστε γιατί προέκυψαν μετά από διαπραγματεύσεις αλλά ε, εκ των υστέρων το να ανακαλύπτουμε ότι πρόκειται για ορισμένα ε, προϊόντα ε, τα οποία είναι σημαντικά για τη μία ή για την άλλη πλευρά, αυτό δεν είναι σωστό. Ε, πρέπει λοιπόν και οι δύο πλευρές να δείξουν ειλικρίνεια και να καταστήσουν σαφές ότι επιθυμούν με απόλυτη διαφάνεια να ορίζουν την κατάσταση που αν το κάνουμε αυτό θα αποκλείεται να συμβούν αυτά που συνέβησαν σήμερα, που βλέπουμε σήμερα. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο, επομένως να δώσω το λόγο στον ε, πρέσβη της Νορβηγίας ε, αν θέλει να κάνει κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, είναι αυτονόητο ότι άκουσα πολύ προσεκτικά όλα όσα είπατε. Και συνήθως ε, τις παλιές μέρες ε, θα λέγαμε θα αναφέρω ε, τόσο ακουμπόθηκα στις αρχές μας, αλλά εφόσον μπορούν να το ακούνε αυτό και απευθείας αναμετάδοση, ήδη το έχουμε καλύψει αυτό. Τώρα, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες επικοδομητικές και φιλικές παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν διαβουλευτήκαμε οι δασμοί στην Ορβηγία αποτελούν ένα του συνολικού προπολογισμού. Η προετοιμασία του συνολικού προπολογισμού είναι ε, μία από τις ε, πιο μυστικές ε, διαδικασίες στις περισσότερες χώρες και υποθέτω ότι αυτό θα ίσχυε και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δασμοί δεν αποτελούν μέρος της δικής σας δημοσιονομικής διαδικασίας καθώς έχετε τελωνιακή ένωση, αλλά για μας είναι μέρος ε, της συνολικής προετοιμασίας του προπολογισμού. Και ε, η κυβέρνηση είχε λάβει αυτή την απόφαση πριν ε, να καταστεί επίσημη. Εγώ ενημέρωσα και την Κομισιόν αλλά και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το τι ετοιμαζόταν και μόλις θα γιατατηθεί η πρόταση θα έπρεπε να το συζητήσουμε επικοδομητικώς. Κάτι που το κάναμε σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο της Κομισιόν, στο επίπεδο των Επιτρόπων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, το θέμα του περιεχομένου αλλά και το γράμμα του νόμου, το βλέπουμε διαφορετικά. Προσπάθησα να εξηγήσω στα εισαγωγικά μου σχόλια. Αν αυτό το δείτε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο του τι έχουμε πετύχει από τότε που ξεκινήσαμε την εφαρμογή των διατάξεων του Αρθροκαλιά. για μένα αυτό δεν είναι προστατευτισμός. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Και για εσά και για μας. Και είπα ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση, προφανώ. Και Έτσι προσπαθώ να εξηγήσω και το τον μέσο αντίκτυπο. Τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία για το επίπεδο των δασμών και τα λοιπά λένε κάτι, αλλά αν δούμε το πραγματικό αντίκτυπο, η δική μας αξιολόγηση είναι ότι θα έχει πραγματικά μελιτέο αντίτυπο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Και για το τυρί. Για Είχαμε δύο γραμμές δασμολογικές από τις 14, δηλαδή δεν είναι ότι αυτό αποτελεί το τέλος της εξαγωγής εταιριού στην Ορβηγία. Το αντίθετο, εδώ μιλάμε για δύο δεσμολογικές γραμμές. Τώρα, για τις ε, ποσοστώσεις. Εμείς ε, χρησιμοποίησαμε μια δημοπρασία, όπως λέμε. Αυτό δεν είναι κάτι σύνηθες ε, στη διεθνή εμπορική πολιτική. Δεν είναι μάλλον κάτι μη σύνηθες. Πολλές χώρες το κάνουν. Και εμείς αυτόν τον τρόπο ακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό. Επίσης αυτό είναι κάτι που συζητείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης ομοτύπων του ΠΟΕ. Θα το αφήσω αυτό κατά μέρο τώρα, αλλά δεν θα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι δική μας εφεύρεση αυτή, γιατί δεν είναι. Και τέλος, για το διάλογο. Ολοκλήρωσα την πρώτη μου παρέμβαση λέγοντας ότι ο ΕΟΧ περιλαμβάνει μηχανισμούς και διατάξει που επιτρέπουν ένα τέτοιο διάλογο. Έκανε συγκεκριμένη αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΟΧ που έλαβε χώρα χθε και προσθέθηκε στο δεύτερο τμήμα αλλά νομίζω ότι στο πλαίσιο των θεσμικών μας σχέσεων όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το διάλογο αυτό. Και με βέβαιος ότι θα το πράξουμε. Και κάτι ακόμη. Εγώ χαίρομαι που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να παρευρεθώ σε αυτή την επιτροπή, να έρθω εδώ να εξηγήσω και να απαντήσω στα θέματα αυτά και θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρεσβευτή και τώρα να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Θα είμαι σύντομο και θα κάνω και τρει παρατηρήσει. Πρώτον, άκουσα τον πρέσβη να λέει ότι οι δεσμοί είναι φυσική ε, απόφαση και φυσική απόρρεια τη διαδικασία για τον νορβηγικό προπολογισμό, όμω οι διεθνεί συμφωνίε είναι και εθνικές αποφάσεις και σε περίπτωση που οι εθνικές αποφάσεις αντίκεινται σε διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να υπερισχύουν οι δεύτερες. Δύο. Όταν ο πρέσβης λέει ότι μας ενημέρωσαν, εγώ να πω ότι υπάρχει διαφορά για την ε, κοινοποίηση μονομερούς απόφασης σε εταίρο και την έναρξη διπραγματεύσεων με τον εταίρο. Και τρίτον, ένας νέος δασμός για τις δύο γραμμές αυτές του τυριού στην Ορβηγία θα είναι 277%. Δηλαδή για για ένα ευρώ τυριού, αυτό θα κοστίζει για τον Νορβηγό εισαγωγέα 278 ευρώ. Αφού εγώ το ονομάζω προστατευτισμό και αυτό το λέω για να ενημερώσω τα μέλη του Κοινοβουλίου. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι και ο πρόεδρος Μορέιρα παρακολουθεί στενά το όλο θέμα και σίγουρα θα θελήσει να δώσει συνέχεια στην όλη συζήτηση. Να ευχαριστήσω πάντως ιδιαίτερα στο πρέσβη και που βρήκατε το χρόνο να έρθετε ως εδώ σήμερα. Να κάνω και εγώ μια παρατήρηση. Είπατε ότι η μετάδοση αυτή μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Και ότι η κυβέρνησή σας ήδη τώρα γνωρίζει αυτά που συζητήθηκαν. Θα χαρώ ιδιαίτερος λοιπόν, λόγω της ζωντανής αναμετάδοσης αυτής της συνεδρίασης, να αλλάξει απόφαση η κυβέρνησή σας. Να κλείσουμε το, τη συζήτηση για το σημείο αυτό και να περάσουμε στο 19 πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά τη Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασίε που αποσκοπούν στη διευκόλυνση διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τη Ένωση στην αγορά τρίτων χωρών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. So this is the first exchange of views. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει ήδη προσελκύσει ιδιαίτερα την προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει οδηγίε που θα ε, διαθετούν τι δημόσιε προμήθειε στην εσωτερική αγορά. Όμω, επιπροσθέτω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά προτείνει ένα νέο εργαλείο το οποίο στόχο έχει να τονώσει τι διαπραγματεύσει και να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στου εμπορικού εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων. Ε, αυτό είναι μια καθοριστική έννοια. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι ανοιχτή σε εταιρείε τρίτων χωρών που θέλουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμού για συμβάσει προμηθειών όμω. Οι ευρωπαϊκέ εταιρείε την χάνουν εσεί μεταχείριση σπανιότατα σε τρίτε χώρε. Γι' αυτό λοιπόν ε, η η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί την πολυετή συμφωνία GPA. Πολλά όμω ακόμη δεν έχουν διαθετηθεί, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να προτείνει κάτι για ένα τέτοιο νέο εργαλείο. Ω εισηγητή για το θέμα αυτό, θα ήθελα να κάνω τι ε, παρατηρήσει μου για το θέμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα ε, κάνει μια παρουσίαση για την πρότασή της και για τα όσα αποφάσισε να προτείνει. εδώ. από τη Γενική Διεύθυνση μπορεί να καλούσε τον κύριο Σλίγκερμαντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να πω ότι η υποβολή τη πρόταση αυτή θεωρήθηκε μέτρο προστατευτισμού, αλλά να σα διαβεβαιώσω για το αντίθετο. Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων, θεωρούμε ότι σε καιρού κρίση και δημοσιονομικών πιέσεων, το περισσότερο εμπόριο είναι λύση. Αυτή είναι η πρώτη μου εναρτήρια παρατήρηση. Η αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή στι προμήθειε από τι τρίτε χώρε κατά το 19% τη αγορά μα. Αυτό δεν ε, ισχύει εδώ στι άλλε χώρε για μα. Υπάρχει δυσκολία πρόσβαση των εταιριών μα, υπάρχει δυσκολία θεμητού ανταγωνισμού σε πολλά μέρη του κόσμου και αυτό δεν είναι απλώς γεγονός, είναι μια πρόκληση που εντείνεται διαρκώς σε όλα ένα περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί κανεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμό εάν δεν έχει τοπική παρουσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αναφερθεί πολλέ φορέ ε, για τέτοιε περιπτώσει και έχουν κατηγορηθεί, αλλά το ίδιο και άλλε οικονομίε. Αυτό οδηγεί σε πολλά προβλήματα. Έλλειψη μόχλευση. Προσπαθούμε να πείσουμε τι διάφορε χώρε να συνάψουν και να προσχωρήσουν στην αναλογική συμφωνία σε επίπεδο και να ανοίξουν τι αγορέ του. Όμω γίνεται το εξή ερώτημα. Ότι εμεί ε, ήδη έχουμε ανοίξει την αγορά μα και δεν έχουμε κάτι να τα Η εσωτερική μα τάξη με τι οδηγίε μα δεν προβλέπουν κάτι για την πρόσβαση τρίτων χωρών. Δεν υπάρχει νομική βάση για τον αποκλεισμό ή ουδήποτε. Αυτό είναι ένα γεγονό χειροπιαστό. Και με αυτό ακριβώ το εργαλείο αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε με την απουσία τέτοιων κανόνων, κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν να έχουν κανόνες αμοιβαιότητας για την πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες, στις αγορές τους. Αλλά ανακεφαλαιώνοντας, στόχος είναι να ανοίξουν οι αγορές και αλλού. Είναι ένα εργαλείο ενθάρρυνσης, παρότρινσης των τρίτων χώρων να ανοίξουν τις αγορές τους. Θέλουμε να προσφέρουμε πρόσθετες ευκαιρίες για εισαγωγές και εξαγωγές, να υπάρχει μόχλευση για τις δικές μας ε, προμηθείες και ίση κανόνες παιχνιδιού, καθώς και συνέπεια. Να ισχύουν αλλού αυτά που ισχύουν και την πρόσβαση στη δική μας αγορά. Η πρόταση τώρα αποτελείται από δύο πυλώνες. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί. Νομικός, οποιαδήποτε ξένη συμμετοχή θα γίνεται αποδεκτή σε διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποκλεισμοί θα είναι η εξαίρεση. Η φορείς ε, προμηθειών θα μπορούν να αποκλείουν κάποιου μετέχοντε σε περιπτώσεις που οι ανάλογοι τομεί προστατεύονται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά και εμεί θα κρίνουμε κατά πόσον υπάρχει ανοιχτή αγορά αλλού ή όχι και έπειτα ο δεύτερο πυλώνα είναι ότι αφού πιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αναλυτική εξέταση του τι συμβαίνει σε άλλε ξένε χώρε και ότι εκεί υπάρχει συστηματικό αποκλεισμό των ευρωπαϊκών εταιριών, τότε να υπάρξει διαβούλευση με τι ε, ε, ενδιαφερόμενε κυβερνήσει και αν δεν βρεθεί λύση, τότε να περιορίσουμε, εφόσον χρειάζεται, την πρόσβαση για άλλα κράτη. Θα υπάρχει στόχευση για συγκεκριμένου διαγωνισμού, όμω θα έχουμε κάποια μέσα πίεση ώστε εφόσον ε, χώρε που αποκλίνουν συστηματικά του δικού μα μετέχοντε, ότι και εμεί μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία. Να ανακεφαλαιώσω τώρα πώ έχει κατάσταση σήμερα. Δεν υπάρχει πολιτική εξωτερικών, ε, εξωτερική πολιτική για, τους δημόσιους, ε, για τις δημόσιες προμήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή και ο κίνδυνος προστατευτισμού από μεμονωμένους φορείς ή κράτη-μέλη όλο ένα και περισσότερο ανακύπτει. Κάποιοι προσπαθούν να προστατεύσουν τι αγορές τους. Στο μέλλον, λοιπόν, νομίζω θα πρέπει να υπάρχει μια εξοδική συνολική εξωτερική πολιτική, ώστε να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στου διεθνεί οργανισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρχουν και περισσότεροι ίσοι κανόνε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Επίτροποι Ντεχούχτ και Μπανιέ στηρίζουν την ε, πρόταση αυτή και θα ήθελα γι' αυτό από την Γενική ε, Διεύθυνση Αγορά να πάρει το λόγο και ο συνάδελφό μου για να με συμπληρώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω λίγε λεπτομέρειε για αυτό που είπε ο συνάδελφο, για την εσωτερική αγορά και τι σχετικέ πτυχέ στην πρόταση αυτή. Από την πλευρά τη εσωτερική αγορά εναρμονίζονται οι έννοιε για την ενδεχόμενο απόρριψη συμμετοχών από του συμβαλόμενου φορεί. Εκεί όπου δεν υπάρχει συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλη χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν κάποια αμοιβαιότητα εδώ. Εφόσον απεκλειστούν συμμετέχοντες, θα μπορεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του σε συμβάσει μέχρι τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα θα μπορούν οι συμβαλόμενοι φορείς να απορρίψουν ξένε συμμετοχέ εφόσον στι χώρε το προελευσή του δεν υπάρχει πρόσβαση για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επιπλέον πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο συμβάσεων που μπορεί να καλυφθούν από αυτή τη διάταξη φτάνει το 40% των συμβάσεων που συνάπτονται ετησίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπόλοιπο 60% θα είναι ανοιχτό στου ε, ξένου επενδυτέ, ε, χάρη στον κανόνα των 5 εκατομμυρίων. Πρόεδρο, ευχαριστώ και του δύο. Και τώρα λοιπόν θα ήθελα να κάνω κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις ε, ως εισηγητής. νομίζω είναι πολύ καλό ότι η Κομισιόν ε, παρουσίασε για άλλη μια φορά την ουσία αυτού του θέματος. Ε, κατά το παρελθόν, δυστυχώς, ε, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση, διότι δεν είχαμε συμφωνήσει οι δύο αρμόδιες επιτροπές για το ποιος ε, είναι, ποια είναι αρμόδια επί της ουσίας και ποια όχι. Τώρα τα βρήκαμε και νομίζω ότι εμείς έχουμε την αρμοδιότητα για τα περισσότερα θέματα αυτά που συζητάμε. Όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες, ε, τους κρατικούς διαγωνισμούς, δημόσιους διαγωνισμούς μάλλον. Ε, υπάρχει βέβαια και κάποια δυνατότητα να συμμετέχει και η Επιτροπή Εμπορίου. Εγώ θα ήμουν ευγνώμων ε, να μην υπάρξει διαφωνία με την Επιτροπή Εμπορίου και όχι διότι δεν αναγνωρίζω το στόχο, αλλά διότι κατά το παρελθόν είχαμε ένα θέμα που ήταν παρεμφερές και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ε, να μην επαναλάβουμε ακριβώς ε, τέτοια θέματα που είχαμε πει και παλαιότερα στην περίπτωση του θέματος του φακέλου ε, Made in που κατασκευάστηκε στην τάδε χώρα. Όπως είπε και η κυρία Μουσκαρντίνη, ε, θα πρέπει να περάσει, να προσπαθήσουμε να περάσει αυτή η έκθεση Μέντε, η οποία δυστυχώ ε, δεν μπορούσε να περάσει στο Συμβούλιο. Και δεύτερον, έχουμε την έκθεση Μουσκαρδίνη, η οποία είχε ε, παραλύσει, είχε αγνοηθεί για δύο χρόνια στο Συμβούλιο και τώρα η Κομισιόν προτείνει να αποσυρθεί πλήρω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί να μην συμβεί με αυτό το θέμα ό,τι συνέβη και στο όλο θέμα γύρω από το Made In. Ε, γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα τι να κάνω εγώ. Καταρχήν πρότεινα ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μας δίνει χρόνο στην Επιτροπή και μας δίνει και κάποιο χρόνο ε, στη διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Εγώ τις προηγούμενες εβδομάδες είχα κάποιες διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους του Συμβουλίου και των κρατών μελών και τελικά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο υπάρχει μία μειοψηφία ε, τροχοπέδη που δεν θέλει να διαπραγματευτεί. Δεν θέλω λοιπόν να ξανασυμβούν, επαναλαμβάνω, αυτά που έγιναν στην περίπτωση Made In. Γι' αυτό λοιπόν θέλω ε, εμείς εδώ στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο με συγχωρείτε, να τα βρούμε το στομό των δυνατών, να ψηφίσουμε και να στείλουμε το θέμα ε, στο Συμβούλιο. Βέβαια πρέπει να έχουμε χρόνο, χρόνο έτσι ώστε να επιτύχουμε συνένεση για αυτό το θέμα και μετά πριν ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας να έχουμε συζητήσει με το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη για να δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κάποια μετακίνηση στο Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν αν υπάρξουν ενδείξεις μετακίνησης στο Συμβούλιο και αυτό το είπα και στην επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να προχωρήσουμε γρηγορότερα, να προτάξουμε την ψηφοφορία, να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Νομίζω όμως ότι ως Κοινοβούλιο εμείς ε, στην όλη η διαδικασία ε, δεν δεσμευόμεθα εφόσον δεν έχουμε ψηφίσει και μπορούμε πολύ πιο εύκολα να ξεκινήσουμε συζητήσεις με τους άλλους θεσμείς από το να έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης στην Ολομέλεια. Γιατί αν κάνουμε το ίδιο λάθος όπως και στο Made in θα βγούμε έξω από τη διαδικασία. Και δεν θέλω να συμβεί αυτό σε αυτό το θέμα, γιατί ξέρω ποια είναι η πλειοψηφία. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί με το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα χαρώ και εγώ αν τις επόμενες εβδομάδες εκμεταλλευτούμε το χρόνο για να διεξάγουμε διαπραγματεύσεις, ε, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και θα ήθελα να φέρω ενδεικτικά. Από το 2004 στον τομέα των κοινοφελών οργανισμών έχουμε τα άρθρα 58 και 59 όπου ε, μπορούν να αποκλειστούν οι ε, αλλοδαποί μετέχοντες ε, σε διαγωνισμούς ε, όταν πρόκειται για κοινοφελείς υπηρεσίες. Κατά την άποψή μου δεν έχει κανένα νόημα να εγκρίνουμε έναν κανονισμό που να καλύπτει το σύνολο των κρατικών προμηθειών. Υπάρχει μια οδηγία η οποία σας είπα ε, για 8 ολόκληρο χρόνια δεν εφαρμόστηκε ούτε μία φορά. Αν λοιπόν το άρθρο ενός κανονισμού δεν έχει εφαρμοστεί για 8 ολόκληρα χρόνια θα πρέπει να σκεφτούμε τι είδους συμπεράσματα πρέπει να εξάγουμε. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάποιες λεπτομέρειες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι να καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το φάκελο και αν το εννοούμε πραγματικά σοβαρά να ξέρουμε ότι έχουμε στα χέρια μας μία σημαντική δύναμη, ένα του. Ε, να δούμε ποια άρθρα είναι σημαντικά ή όχι, η ε, τοπική αυτοδιοίκηση ε, να προσπαθήσει ε, να μπει στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν είναι τόσο καθοριστικό όσο τα άρθρα 8 και 10. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προτείνω στους σκιώδεις εισηγητές την ε, επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο να συναντηθούμε, να δούμε τι πιστεύουν εκείνοι και από κοινού να δούμε και τι συζητήσεις θέλουμε να έχουμε. Ε, εγώ πρέπει να σας πω ότι ό,τι επιθυμίες έχουν οι σκιώδεις ηγητές θα τις λάβω υπόψη μου γιατί ενδιαφέρομαι να υπάρξει ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο γιατί αλλιώς θα συμβεί αυτό που έγινε με την περίπτωση Made In. Επίσης αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συζητήσουμε με τις χώρες εκείνες που αυτή τη στιγμή μπλοκάρουν την όλη υπόθεση στο Συμβούλιο. Γιατί αν δεν κατορθώσουμε σε πρώτη ανάγνωση να βρούμε κάποια λύση μαζί με το Συμβούλιο, ε, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Να κλείσουμε την πρώτη ανάγνωση, να πάμε στον τρίλογο και ε, σε δεύτερη ανάγνωση ε, να ολοκληρώσουμε το όλο θέμα πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Άρα δηλαδή ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και μετά ενδεχομένως ε, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου να υπάρξει, ε, να κλείσει το θέμα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχω κατά νου. Αλλά σας λέω για άλλη μια φορά, αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να μην πάθουμε αυτό που πάθαμε με το Made in. Να επιτύχουμε ευρεία συμφωνία στο Συμβούλιο και να προχωρήσουμε στο Κοινοβούλιο και να προχωρήσουμε στο Συμβούλιο. Uh, Um, να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους, πρώτα στον συνάδελφος Σούστα για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να πω ότι δεχόμαστε την ε, πρόσκληση να βρεθούμε σύντομα στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμη μια συνεδρία των σχεδόν εισηγητών για να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Δεύτερον, επί της ουσίας, είναι σαφές ότι εμείς ε, συμφωνούμε με το πώς παρουσιάζεται αυτή η πρόταση κανονισμού, γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο τομέας ε, των ε, δημοσίων διαγωνισμών και πόσο ελλειπές είναι το σύστημα των διεθνών κανόνων και γιατί οι αναδυόμενες ε, χώρες, ε, ίσως θα ήταν ε, καλύτερα βέβαια να βρούμε μια άλλη ορολογία, να μην τις αποκαλούμε αναδυόμενες χώρες, γιατί είναι εδώ και τόσο καιρό αναδυόμενες, ενώ είναι τελικά ανταγωνίστριες, πληρώ ανταγωνίστριες της ευρωπαϊκής μας οικονομίας και δεν έχουν λοιπόν προσχωρήσει στη συμφωνία GPA και εμείς ε, βλέπουμε εδώ να μην έχουμε ένα διεθνές πλαίσιο κανόνων που να μας προστατεύει και να δημιουργεί συνθήκες αμοιβαιότητας. Ήταν ε, λοιπόν δεν ευπρόσδεκτη μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε ορισμένα συγκεκριμένα άρθρα αυτού του κανονισμού. Αναφέρω το άρθρο 6, το 8, το 10. Αυτά θα πρέπει να εξεταστούν εις βάθος και νομίζω ότι θα είναι επίσης σωστό να, να έχει καλυφθεί όλα η, η ύλη που αυτή τη στιγμή σήμερα προσδιορίζεται με τις τρεις οδηγίες που νομίζω συζητούνται στην Επιτροπή ΙΜΚΟ σήμερα και πολλές φορές ε, ε, έχει γνωμοδοτήσει και ΙΝΤΑ επ' αυτών. Επομένως, ε, θα ήθελα να διαπιστώσω ότι ε, υπάρχει μια οριζόντια συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε και λίγο περαιτέρω όχι μόνο για τους γιονισμούς που ψευρούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ που είναι το 7% των ε, συνολικών ε, γιονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε και περαιτέρω εις βάθος ε, για το τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που έχουμε εμφανιστεί κάτω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ορισμένου τομεί λαμβάνεται υπόψη ότι το σύστημα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ε, δεν συμμετέχει πολύ συχνά σε αυτές τις διαδικασίες άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό επί της ουσίας τώρα σε σχέση με πιο τυπικά πράγματα, σε σχέση με τις ανησυχίες ε, που ο εισηγητής και πρόεδρος μας Εξεδηλώσε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι η σοφροσύνη στην περίπτωση αυτή είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να ξεφύγει, να διαφύγει για να επιλύσουμε ένα κυρίως πολιτικό ζήτημα. Το πρώτο δίδαγμα που έρχεται από το ΜΕΙΤ είναι ακριβώς αυτό, να μην επαναλάβουμε αυτό το, αυτή την εμπειρία, δηλαδή να μην ε, βιαστούμε εμεί, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι θέλουν το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Τι θέλει η Κομισιόν, το καταλάβαμε. Διαφορετικά θα έχει παρουσιάσει η νομοθετική πρόταση. Τώρα, από την πλευρά του Συμβουλίου, πόσο αποδεκτή είναι η πρόταση αυτή, το γνωρίζουμε αυτό. Σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται το Συμβούλιο και υποθέτουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση. Όμως εγώ πιστεύω ότι αν έτσι έχουν τα πράγματα θα μπορούσαμε και από τώρα να αναστείλουμε τις εργασίες μας. Όμως αντίθετα πιστεύω ότι το καθήκον της Κομισιόν αφενός και του Κοινοβουλίου αφετέρου, θα έλεγα και δύο από κοινού, με το πραγματικό κοινοτικό κεκτημένο, με το πραγματικό σύστημα των θεσμικών σχέσεων που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις Ευρωπαϊκές Ένωσης είναι μια ισχυρή σχέση Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Και έτσι εμείς έχουμε και το καθήκον μάλιστα να εργαστούμε πλάι στο Συμβούλιο. Γιατί το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό, να κατανοήσουμε πολιτικά αν το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται πώς ενώπιον ε, αναδειμένων διχωρών, όχι αναδυόμενων, ε, γιατί όσες αναδύονται αυτή τη στιγμή, εντάξει, να τους ε, συμπεριφερθεί ευνοϊκά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τις ενθαρρύνουμε, να σεβαστούν ανθρώπινα δικαιώματα, να εκδημοκρατιστούν, να υπάρχει ουσιαστικά μια ανταπόκριση των προσπαθειών τους να αναδυθούν, αλλά όταν έχουν ήδη αναδυθεί χρησιμοποιούν ε, αυτή την ε, έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και προβαίνουν σε θέμα του ανταγωνισμού και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Οπότε λοιπόν δεν έχει πλέον νόημα να επικαλούνται ότι είναι ακόμη αναπτυσσόμενος για να μπορούν να αιτιολογούν όλες συγκεκριμένες συμπεριφορές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Όμως θέλω να σημειώσω και κλείνω πρόεδρε εδώ ότι οι ανησυχίε σου σε σχέση με το να μην επαναληφθεί όλη αυτή η ιστορία με το Made In, ε, βλέπουμε εδώ να υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ της υπόθεσης Made In και της υπόθεσης που συζητούμε εδώ, γιατί οι παλιές οδηγίες για τους δημοσίους αγωνισμούς και αναφέρομαι στη σχέση μεταξύ της δικής μας Επιτροπής με την Επιτροπή Εμπορίου. Υπήρχαν λοιπόν, υπήρχε στις παλιές οδηγίες μια διάταξη για την αμοιβαιότητα, ενώ σήμερα αυτή η διάταξη έχει φερεθεί από τις νέες οδηγίες για τα δημόσια έργα αν ε, αυτό το οποίο εμείς το ψηφίσαμε ήδη και σε λίγο θα ψηφίσει σε λίγους μήνες η Επιτροπή οικογένεια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, χωρίς να υπάρχει μία διάταξη σαν αυτή, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία, η Ευρώπη κάνει ένα βήμα πίσω στο σύστημά της, ε, στο να υπερασπίζεται και να προστατεύει την αμοιβαιότητα. Γι' αυτό λοιπόν ε, υπήρξαν ε, τροποποιήσεις στις οδηγίες ε, για τις παραχωρήσεις. Το κάναμε αυτό γιατί εδώ υπάρχει κίνδυνος νομοθετικής ψήφου. Ο κανονισμός αυτός, αυτή η οδηγία δηλαδή που θα καλύψει αυτός ο κανονισμός από γενική σκοπιά, αλλά αν δεν προχωρήσει αυτός ο κανονισμός, τότε εμείς αντίθετα με το τι ισχύει σήμερα, σε λίγους μήνες θα μπορούσαμε να βρεθούμε στον κίνδυνο να μην έχουμε ένα σύστημα προστασίας. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε τις τροπολογίες εκείνο το βήμα και πρέπει να διαπιστώσουμε δυστυχώς ότι ε, αυτό το ζήτημα δεν έγινε έπαρξη κατανοητό στο βήμα της ΣΥΝΤΑ. Έτσι λοιπόν, να προχωρήσει να μένει η έκθεση αυτή, αλλά ταυτόχρονα έχουμε την αίσθηση ότι δεν προχωράω ο στην ΙΜΚΟ την νομοθεσία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ω τροπολογία. Γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα έχουμε ούτε αυτόν τον κανονισμό και θα έχουμε οδηγίε που θα βοηθήσουν την είσοδο του οποιοδήποτε και με οποιασδήποτε συνθήκες στους ευρωπαϊκούς δημοσιογονισμούς. Κάτι που θέλαμε εμείς να αποφύγουμε. Να απαγορεύσουμε και νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια του χρόνου. Εμείς είμαστε υπέρ οποιασδήποτε μεσολάβησης, αλλά εδώ διαφέρει η κατάσταση από το ΜΕΝΤΙΝ, γιατί εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε καθοδόν συστήματα προστασίας του δικού μας συστήματος ε, που αποτελούσε εγγύηση για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Ε, ε, Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Καζάκα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, και εγώ είμαι της άποψης ότι αυτή η συζήτηση είναι άκρα σημασία και ιδιαίτερα επίκαιρη. Καλωσορίζω την ιδέα του εισηγητή μας να οργανωθεί συνάντηση μεταξύ του ιδίου και των σχεδόν εισηγητών ώστε να καταρτήσουμε μια ενιαία στρατηγική για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίκαιρο λοιπόν είναι και πολύ σημαντικό, είναι εξέχουσα σημασία αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τι δημοσιονομικέ αποφάσει. Βεβαίω, εδώ μιλάμε για δημόσιε προμήθειε που είναι ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα και σημαντικά θέματα για την εμπορική μα πολιτική. Για τον εξή βασικό λόγο. Μιλάμε για κυβερνητικέ επί τη ουσία συμβάσει. Οι συμβάσει αυτέ ε, καλύπτονται και πληρώνονται από του φορολογουμένου. Στην περίπτωση αυτή όταν εμπλέκονται ο δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο και να πετύχουμε δύο βασικούς στόχου που κάποιε φορέ είναι αντιφατικοί. Πρώτα απ' όλα, αναζητούμε την ε, πλέον ευνοϊκή τιμή για τον ε, φορολογούμενο και έπειτα θέλουμε να στηρίξουμε την εγχώρια οικονομία, την εγχώρια βιομηχανία. Λόγω του δι του αυτού στόχου και παρόλο που είναι θεμητή, κάποιες φορές έχουμε καταλήξει σε ακραίες καταστάσεις. Διότι κάποιες φορές πετύχαμε τους στόχους μας με φτηνότερες τιμές, αλλά με κακή ποιότητα. Ή έχουν ε, δημιουργηθεί εθνικά μονοπόλια και έτσι πλήττεται το ελεύθερο εμπόριο. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω, για τον οποίο πιστεύω ότι η συζήτηση που θα πρέπει να γίνει σήμερα δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί στο εάν είμαστε υπέρ ή κατά της αμοιβαιότητας ή εάν είμαστε υπέρ ή κατά του ελεύθερου εμπορίου ή του προστατευτισμού. Ως φιλελεύθερος και δημοκράτης θα ήθελα να δώσουμε έμφαση σε άλλα σημαντικότερα ζητήματα. Δηλαδή, ποια είναι η προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας. Με ποιο τρόπο η εμπορική μας εταιρεία από τρίτες χώρες θα ανοίξουν περισσότερο τις αγορές τους εμάς. Και πάνω απ' όλα, ποιο είναι το σύνολο εργαλείων που θα πρέπει να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιδιώξει του στόχου αυτού στο διεθνέ προσκήνιο και στι διεθνεί εμπορικέ διαπραγματεύσει. Νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να διέπει ολόκληρη την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρόταση που σήμερα εξετάζουμε. Ιδίω πώ οι αγορέ των τρίτων χωρών θα μπορέσουν να ανοίξουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο επίπεδο των δημόσιων προμηθειών. Βεβαίως η συμφωνία για τις κυβερνητικές συμβάσεις στον ΠΟΕ υπάρχει. Βεβαίως είναι συμβαλόμενο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ανέφερε εδώ ο συνάδελφος ότι υπάρχουν μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες που δεν έχουν συμπληθεί στη συμφωνία αυτή και δεν έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία μαζί τους ε, για σχέσεις ελεύθερου εμπορίου. Λόγω χάρη με την Κίνα. Έτσι λοιπόν, πολλά είναι τα ζητήματα που ανακύπτουν. Πολλά τα προβλήματα. Η πολιτική για τις δημόσιες προμήθειες, η εξωτερική μας δηλαδή πολιτική για τις δημόσιες προμήθειες, έχει αδυναμίες. Διότι από τη μια ανοίγουμε την αγορά μας για τις εταιρείε τρίτων χωρών, αλλά το ίδιο δεν κάνουν και οι εταίροι μας. Και δεν έχουμε και τη δυνατότητα να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Ακριβώς, διότι δεν υπάρχει ένα σχετικό εργαλείο, ένα κουτί εργαλείων που να το εμπιστευόμαστε, που να βρίσκεται στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θα στηρίξω ως αποτείνονται στο σχέδιο κανονισμού πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 8 και 10 όπου οι προκαταρκτικές μελέτες και οι διαβουλεύσεις προαπαιτούνται, οπότε στην περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μπορούν να υιοθετηθούν μόνο μερή, μάλλον μέτρα αμοιβαιότητας. Φυσικά κάποια πράγματα πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο, όπως η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 6 Κατά την άποψή μου και με κάθε ειλικρίνεια, αυτό κάπως αντιφάσκει με την πρώτη διαδικασία που προτείνεται και δεν νομίζω ότι μπορούν να συνεπάρχουν στο ίδιο έγγραφο, διότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις. Λόγου χάρη, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίσει διαδικασία διαβουλεύσεων ή ε, εκπονήσει μελέτη κατά της Βραζιλίας βάσει των διαδικασιών που προβλέπουν τα άρθρα 8 και 10 και ταυτόχρονα απορρίψει προσφορά σε διαγωνισμό για δημόσια προμήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφορά της ε, Βραζιλίας, τότε η πρώτη διαδικασία που έχει ξεκινήσει με την βραζιλιανική πλευρά αντιφάσκει με τη δεύτερη. Και αυτό που μα απασχολεί είναι αν τελικά στην πραγματικότητα θα υπάρξει άνοιγμα τη βραζιλιανική αγορά ή κάποια άλλη τρίτη χώρα τέλο πάντων. Ή μήπω συμβεί το ακριβώ αντίθετο. Δηλαδή, μήπω έχουμε αντίπεινα, οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Ε, είναι η αντίδραση που προκαλέσουμε. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε αυτό τον πρωταρχικό στόχο, το ακριβω αντιθετο δηλαδη μηπω εχουμε αντιπεινα οφθαλμον αντι οφθαλμου ειναι η αντιδραση που προκαλεσουμε πρεπει λοιπον να επιδιωξουμε αυτο το πρωταρχικο στοχο το ανοιγμα των αγορών των τρίτων χωρών και όχι περαιτέρω προστασία του. Μην ξεχνάμε ποτέ αυτή την ιδέα κατά τη συζήτηση τη πρόταση αυτή για το σχέδιο κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμεί πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζαντό εκ μέρους των ε, Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτό το δόγμα ακολουθεί και το δόγμα άλλων οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες και βλέπουμε ε, στις κλασικές οδηγίες ε, την ενσωμάτωση κοινωνικο-περιβαλλοντικών κριτηρίων και αυτό είναι κάτι καλό. Αλλά εμένα με εντυπωσίασε κάπως ε, αυτή η πρόταση κανονισμού στο σημερινό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο κρίσης οικονομικής, βαθιάς οικονομικής ύφεσης, σε ένα πλαίσιο βιομηχανοποίησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή να μπορούμε έτσι απλώς ε, να λέμε ε, ότι Αφρικανική Σύμβαση είναι κάτι κακό, αναγκαστικά αυτό με εκπλήσει. Δεν ε, έχουμε ε, κάποια διδάγματα εμπορικής πολιτικής, ε, να μάθουμε από τις ΗΠΑ σε αυτό το πλαίσιο της κρίσης. Γιατί αν εγώ άκουσα ορθά τους στόχους που μας παρουσίασε η Κομισιόν, μας είπε ότι υπάρχει ένα εργαλείο ίσως με αντίπεινα στις δημόσιες συμβάσεις μας έναντι μιας σειράς χωρών που δεν θα είχαν ανοίξει αρκετά την αγορά των δημοσίων συμβάσεων στις δικές μας επιχειρήσεις αλλά να υπενθυμίσω ότι ο αριθμό αυτών και των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Συμβάσεων που έχουν κερδίσει ξένες επιχειρήσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρός. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει εξέλιξη, αλλά α ε, σημειώσουμε ότι πολύ συχνά τα κράτη, οι συλλογικότητε που έχουν σε μια διαδικασία ε, δημοσίων συμβάσεων θέτουν ε, αρκετά τεχνικά κριτηρία για να διασφαλίσουν ότι πολύ συχνά μια κρατική επιχείρηση θα πάρει τη σύμβαση. Όμως ε, να ότι στην Πολωνία ε, κερδίθηκε από την Κίνα ε, μια προσφορά και θα μπορούσαμε ίσως να δούμε πολλαπλασιασμό τέτοιων περιπτώσεων. Όμως ε, είμαστε σε μια λογία σαν ανοίξουμε περαιτέρω τις ε, δημόσιες συμβάσεις των άλλων κρατών. Ε, υπάρχουν η Κίνα και άλλα κράτη που είναι κλειστά θα λέγαμε και από αυτή τη σκοπιά το θέμα της αμοιβαιότητας είναι νόμιμο. Όμως ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην μπερδεύουμε κράτη όπως η Κίνα που ίσως δεν είναι αναπτυγμένες χώρες από τη σκοπιά του εισοδήματος των κατοίκων, αλλά είναι σίγουρα μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις. Υπάρχουν και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Ο απολογισμός ε, της πολιτικής απελευθέρωσης των χωρών αυτών είναι ότι τουλάχιστον έχουν χάσει με κάποια εργαλεία της δημόσιας πολιτικής γιατί δεν έχουν πλέον δασμούς τελωνιακούς και το εσωτερικό σύστημα φορολόγησης είναι πάρα πολύ αδύναμο. Και αυτό που θα μπορούσαμε δυνάμει να πούμε επίσης ότι δεν έχουν πλέον δημοσιονομικά έσοδα, αλλά το εργαλείο αυτό, το δημόσιο, δεν θα είναι πλέον ένα εργαλείο που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει την αναπτυξιακή της πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτούμε τι είδου ε, αγορές θέλουμε να ανοίξουμε. Αλλά αυτό που εγώ έλεγα και επαναλάμβανα πάντα είναι ότι όσοι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Βραζιλία, άλλε χώρες έχουν εμπορικές πολιτικές που, ε, που μπορούν να ερμηνευθούν ως ξεκάθαρες εμπορικές βιομηχανικές πολιτικές, τελικά η ευρωπαϊκή ε, λογική ε, είναι κακή. Δηλαδή μένουμε σε μία λογική ότι το άνοιγμα θα χρησιμεύσει στη δική μας βιομηχανία και όχι ότι τα δικά μας εργαλεία ε, της πολιτικής θα πρέπει να εξυπηρετήσουν μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Και εγώ θεωρώ ότι σήμερα είμαι υπέρ της λογικής του ανοίγματο, να μπέρξει αμοιβαίο άνοιγμα και όχι σε μια λογική να πούμε ποια είναι τα δικά μας συμφέροντα σε περίοδο κρίσης, ποια είναι τα επιθετικά μας συμφέροντα στην παγκόσμια οικονομία του 21ου αιώνα. Να μην θέτουμε την ερώτηση αυτή. Και να πούμε ότι με κράτη που έχουν μικρό οικονομικό περιθώριο και να λέμε ότι ε, όταν ε, μιλάμε για κάτι που ανταποκρίνεται στο 20% του ΕΠ και αυτό δεν ε, είναι τμήμα της πολιτικής τους, αυτό πραγματικά με εκπλήσει, δηλαδή να απορρίπτουμε κάτι τέτοιο λόγω δογματισμού. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν με την πρόταση κανονισμού. Θεωρούμε πάντοτε ότι θα πρέπει οι δημόσιες συμβάσεις να εξυπηρετούν την ευρωπαϊκή οικονομία όχι με προστατευτικό τρόπο, αλλά ε, λέμε ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία προστατευτισμού. Είχαμε τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για το κινέζικο ντάμπινγκ την περασμένη εβδομάδα. Θα μου πείτε, α, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό τον κανονισμό τον οποίο μιλάνε. Όμω, εν μέρει έχει να κάνει. Όταν η Ευρώπη είναι μέλο ε, του ΠΟΕ με την Ιαπωνία κατά του Καναδά ε, και καταφέρεται σε μια ε, πολιτική που έχει δώσει γεωγραφική προτίμηση, δηλαδή εμείς ε, καταπολεμούμε τη δυνατότητα του Καναδά ε, και λέμε ότι προτιμώ με πραγματικά κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας να ευνοήσω κάποιες επιχειρήσεις τοπικά, μικρές και μισές επιχειρήσεις. Και εγώ δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι ανόητο στον κόσμο που ζούμε. Και η Κομισιόν να απορρίπτει έτσι λίγο. Α, οι Αμερικανοί κάνουν Αμερικανικέ συμβάσει, ε, τίποτα δεν έχω καταλάβει την οικονομία. Εγώ αυτό το βρίσκω πραγματικά εντυπωσιακό. Νομίζω ότι τουλάχιστον ε, θα έπρεπε κάποια στιγμή και ελπίζω ο Ντανιέλ ε, ω ηγητή να πάει τη συζήτηση αυτή και στου κόλπου τη Επιτροπή Ελπίζω λοιπόν να κάνουμε μία συζήτηση για να δούμε αν στον κόσμο με τον οποίο ζούμε σήμερα είναι οι Αμερικανοί που έχουν μεγάλη βιομηχανική πολιτική και οι Κινέζοι που έχουν μεγάλη βιομηχανική πολιτική. Βέβαια, αμφισβητούμε κάποια εργαλεία ντάμπινγκ, αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη βούληση. Εμεί δεν έχουμε τη βούληση αυτή, ότι μα ενδιαφέρει η αμοιβαιότητα των ελεύθερων συλλογών και το μεγάλο άνοιγμα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει πολύ σοβαρά να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα στο ιστορικό τη Επιτροπή μα και Ελπίζω να το κάνεις εσύ, Ντανιέλ Κασπαρή, ως συζητητής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάλφο, στη συνάλφα Μακλάκη, εκ μέρου των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά και πρόεδρε. Είστε σήμερα και πρόεδρος. Ε, δημόσιε συμβάσει είναι ιδιαίτερα σημαντικές ε, ως ποσοστό στο ΑΕΠ μα. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η έκθεση. Ε, αυτή τη στιγμή βέβαια βιώνουμε μια οικονομική κρίση και γι' αυτό πρέπει να προσφέρουμε πραγματική αξία, να δώσουμε την πραγματική αξία στο χρήμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ σήμερα η Κομισιόν και έχει ήδη μιλήσει για την εισαγωγή συγκεκριμένων προτάσεων και ίσως μπορεί να μας απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις που θέλω να υποβάλω εγώ σήμερα, έτσι ώστε να κατανοήσω και εγώ καλύτερα τους στόχους και την κατεύθυνση αυτής της πρότασης ε, και ποια κατεύθυνση θα ακολουθηθεί πιο συγκεκριμένα. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις που είχατε με επιχειρήσεις και με διάφορα κράτη-μέλη. Είπατε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για αυτή τη νομοθετική πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ε, τους τομείς ε, και τα κράτη-μέλη στα οποία αναφέρεστε στη διαδικασία διαβουλεύσεων. Επίσης θα ήθελα να ακούσω λιγάκι το σκεπτικό σας τι συνέβη όταν η Επιτροπή Αξιολόγηση Αντικτύπων υπέβαλε τη δική της την έκθεση, κυρίως ε, όσον αφορά τις ε, τρίτες χώρες ε, και την αγορά των δημόσιων διαγωνισμών. Τα δικά σας, οι δικές σας απόψεις επ' αυτού του θέματος. Επίσης, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ακούσω κάποιες μελέτες από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο οι οποίοι ανησυχούν όσον αφορά το αυξανόμενο κόστος. Μιλάνε για περίπου 60% αύξηση του κόστους για κάποιες συμβάσεις ε, σε αυτόν τον τομέα. Βεβαίως ε, όλοι ε, θέλουν να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα δημόσιων διαγωνισμών που να κοσταλγούν σωστά το χρήμα. Ίσως ε, νομίζω ορισμένα κρατημέλη έχουν αμφιβολίες για την ελεύθερη μετακίνηση των αγαθών που αυτό, αυτή μπορεί να ε, παρεμποδιστεί από την πρόταση τη δική μας. Εσείς τι πιστεύετε, υπάρχει εκεί πρόβλημα και υπάρχει κάποια νομική συμβουλή που μπορείτε να μας δώσετε για να διευκρινιστεί. Επίσης, ε, θα ήθελα να ρωτήσω ε, ποιες είναι οι συμβουλές της νομικής υπηρεσίας ε, και από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Γιατί ανησυχούμε συνεχώς για το αυξανόμενο εμπόριο, για τις εξωτερικές σχέσεις. Αυτά θα έρθουν έγκαιρα για να βοηθήσουν ή όχι κατά τη δική σας άποψη. Ίσως μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτές τις ε, ερωτήσεις. Και εμείς ευχαριστούμε. Έχω άλλους δύο συναδέλφους ε, στον κατάλογό μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σόλτς. Εγώ θα σηκώσει το χέρι μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα ε, πρόεδρε και να συμφωνήσω μαζί σας. Και εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Χρειαζόμαστε κυρίως ε, μία συνεννόηση για τους μακροπρόθεσμους στόχους αυτής της διαδικασίας. Εφόσον μιλάμε για διείσδυση στις αγορές, ε, τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα και τις τελευταίες εβδομάδες, ε, δηλαδή πώς συμβάζονται αυτά με τους ε, επενδυτές ε, δεν φτάνουμε δηλαδή εδώ λιγάκι και στο θέμα των επενδύσεων. Μέχρι ποιο βαθμού ανοίγουμε τις αγορές εάν σε ορισμένες περιοχές και χώρες η οικονομική εξέλιξη είναι τελείως διαφορετική. Εχθές και σήμερα, εχθές, εχθές ψηφίσαμε Σήμερα, σήμερα, με συγχωρείτε, χθε συζητήσαμε και σήμερα ψηφίσαμε για την Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών με το Περού και την Κολομβία. Τι σημαίνει για την κατάσταση σε αυτές τις χώρες, για τους απασχολούμενους σε αυτές τις χώρες, το να συμμετέχουμε εμείς σε διαγωνισμούς τους. Αυτό δηλαδή θα βελτιώσει την κατάσταση, θα τους προσφέρει κάτι. Υπάρχουν ε, πολλά ερωτήματα και σε άλλες υποθέσεις, σε άλλους τομείς που σχετίζονται όμως με το δικό μας. Και αυτά που είπατε εσείς ε, είναι συμβατά ε, με αυτά ε, που έχουμε συζητήσει για θέματα εξωτερικού εμπορίου. Για άλλη μια φορά λοιπόν αυτό που με ενδιαφέρει είναι η συμβατότητα των εργαλείων, η κατεύθυνση του εμπορίου. Αυτά να εξεταστούν. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με συγκεκριμένα κεφάλαια έχουν να κάνουν με κεφάλαια στις ε, συμφωνίες εμπορικών ανταλλαγών, ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών που έχουν ήδη υπογραφεί. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι η κυρία Γενίκη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή συζητάμε για αυτή την πρόταση ε, μεσούσης της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση αν έχουμε την τάση ότι ανοίγουμε απέναντι σε σένα όσο ανοίγεις και εσύ απέναντι σε μένα και αυτό το έχουμε αναγάγει σε αρχή οικονομικής συνεργασίας. Εγώ δεν ξέρω, αμφιβάλλω επ' αυτού γιατί αυτό έχει ε, προκλήσεις βιομηχανικές, οικολογικές, ε, κοινωνικές, πάρα πολλές. Έχει πολλές συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο να συνεργαστούμε με την ΙΜΚΟ στο θέμα της ψηφορίας και στο πού κατευθύνεται όλο αυτό το εργαλείο. Τρεις ακόμη έχουν ζητήσει το λόγο από τους συναδέλφους. Ο Κρίστοφερ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ασκήσω κριτική και νομίζω ότι έχω τέσσερα σχόλια. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δημοσίες συμβάσεις, ε, για να ξεκινήσουμε. Ποιος ο λόγος για να μου για τις δημοσίες συμβάσεις. Όπως το ερμηνεύω εγώ, είναι σημαντικό να έχουμε μία δίκαιη διαδικασία μεταξύ όσων ανταγωνίζονται για κυβερνητικά χρήματα, όχι χάρες, όχι διαφθορά. Δεύτερον, να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα για τα λιγότερα χρήματα. Γιατί θέλουμε αξία για τα χρήματα των φορολογουμένων και αυτό νομίζω ότι είναι σε ακόμη λόγος και ειλικρινά πιστεύω ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ δυσνόητη. Το ακούσαμε και νομίζω ότι έντιμε η Κομισιόν ε, το είπε ότι αποκαλείται προστατευτισμός. Κάποιος που το έκανε νομίζω ότι ήταν ε, ο κύριος Λαμή από τον ΠΟΕ και πρώην επίτροπος είπε ότι εμφανίζεται ένας προστατευτισμός και αυτό το με κάνει υπερήφανο. Και επίση πιστεύω, ακούω από την Κομισιόν, σαν διαβεβαίωση ότι το 60% των αγορών θα παραμείνουν ανοιχτέ. <laughs> Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάπως προκλητικό όταν ε, λέμε ότι ε, το 60% των αγορών θα παραμείνει ανοιχτό. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι κακό αν δούμε και την οικονομική συγκυρία, την παγκόσμια οικονομική κρίση και το ότι έχουμε παγκόσμια αναζήτηση νέου προστατευτισμού. Νομίζω ότι ήταν κακό να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Τώρα, κάτι ακόμη. Πιστεύω ότι από αυστηρό ευρωπαϊκή σκοπιά, όταν εμεί είμαστε σε οικονομική κρίση, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Γιατί ότι δεν θυμάμαι πόσες φορές ε, άκουσα τον πρόεδρο Μπαρόσο να ε, μιλά για το πόσα χρήματα θα δαπανίσουμε για να επενδύσουμε στο δημόσιο τομέα, για να δώσουμε κίνητρα στην οικονομία και δεν μπορώ να δω κανέναν άλλο τρόπο με τον οποίο θα έφυγε αυτή η ροποθυσία, θα έρθει μια τέτοια όθηση, απλώ θα την καθιστούσε πιο ακριβή. Αν αποκλείσουμε κατά κάποιο τρόπο τις ε, φθηνές προσφορές, τότε θα υπάρξει κόστος. Οι κυβερνητικές επενδύσεις θα είναι πιο ακριβές και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να το πράξουμε αυτό οικονομικά. Και δεν είναι ένα θέμα μόνο για τους υπουργού ε, αρμόδιους για το εμπόριο. Ελπίζω και οι υπουργοί οικονομικών να, ε, να το διερευνήσουν αυτό το θέμα και να ρωτηθούν ποιε θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειε αυτού αν αποφάσισαν να το κάνουν οι περιφέρειες, ποιο θα ήταν το οικονομικό κόστος. Και αναγνωρίζω, όπως λέει η Κομισιόν, ότι αυτή είναι μια απόπειρα να ανοίξουμε τις αγορές αλλού. Δηλαδή ότι υπάρχουν και κάποια θετική σκοπή. Όμως ανησυχώ ότι τελικά δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρετε, δεν ε, είναι ως συνέπεια μην κάνουμε να σκεφτούμε πώς θα ανοίξουμε ε, τις ε, ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις. Και η απάντηση από την Κίνα πιθανότατα δεν θα ήταν «Α, εντάξει, κάναμε λάθος, ας ανοιχθούμε». Νομίζω το αντίθετο θα δούμε. Άκουσα την Κομισιόν. Μπορεί κάτι να παρανόησα, αλλά δεν νομίζω να παρανόησα γιατί συχνά γιατί ε, ξέρουμε ότι τα κράτη προσπαθούν ε, να στρεβλώσουν τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών και μπορούμε, αν εναρμονίσουμε, να σταματήσουμε τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς είναι σαν ε, ε, να τις πρόχνουν την Κομισιόν τα κράτη-μέλη να κάνει κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή την Κομισιόν θέλω εγώ. Αν τα κράτη-μέλη έκαναν κάτι στον τομέα αυτό, ουσιαστικά που θα κατακρεμάτιζε την ε, εσωτερική αγορά, τότε εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να υπερασπιστεί τη συνθήκη και να προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη των κρατών μελών, αλλά να επιβάλλει τους κανόνες όχι να επιτραέψει να την εκφοβήσουν τα κράτη-μέλη για να στεγαγεί κάτι, έτσι όπως θέλουν αυτά. Λοιπόν, χάσαμε μια ερώτηση. Χώρες συγκεκριμένου ε, συστήματος ε, προτιμήσεων. Ναι, ναι, έχουμε ε, αυτή τη διαδικασία. εντάξει, αλλά δεν το πίστευουμε, αλλά βλέπουμε ότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αποτελέσματα από τα γραμμάτια και αν δεν πιστεύουμε σε αυτό ίσως θα έπρεπε να το καταργήσουμε, θα ήταν λυπηρό. Αλλά ελπίζω να αποκλείονται οι χώρες GPA, ίσως να μπορεί να μας διαφωτίσει η Κομισιόν. Ε, Ευχαριστώ. Η έκθεση μου κατά την η έκθεση αυτή, κατά την άποψή μου, έχει καθυστερήσει πολύ. Θα έπρεπε να την έχουμε πολύ νωρίτερα. Και δράτω με τι ευκαιρίε για να πω ότι είναι καλύτερα να καθυστερήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο προτού εγκριθεί. Διότι αν δεν καταρτήσουμε ένα εμπόριο νόμιμο, θεμητό και ε, δίκαιο, με δίκαιες συναλλαγές, ο προστατευτισμός των κρατών θα ε, κυριαρχήσει. Ήδη οι προστατευτικέ τάσει των περισσότερων κρατών είναι πολύ ισχυρέ και η μόνη απόκριση στον προστατευτισμό αυτό τη επαναδίπλωση, τον παλιόγνωστο προστατευτισμό, είναι η απάντηση με ένα δίκαιο και ισότιμο εμπόριο που να βασίζεται σε τρεις αρχές, την αμοιβαιότητα, την ισορροπία και το σεβασμό των ε, διεθνών ε, προδιαγραφών όπως έχουν προκύψει μέσα από διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Ε, με πρώτες τις αναδυόμενες χώρες που πρέπει να σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία και την ε, διανοητική. Λέγοντας αμοιβαιότητα, εννοώ ε, αμοιβαιότητα με κεφαλαίο και για τις χώρες που έχουν αναδυθεί και για τις αναδυόμενες. Αυτές έχω στο μυαλό μου. Τώρα για τις χώρες ε, τις λιγότερο ανεπτυγμένε, ε, όπως λέγονται ή τις φτωχέ απλώς, τις μη ανεπτυγμένε, εκεί θα πρέπει να υπάρξει κάποια ε, συμμετρία που να εφαρμοστεί στα μέτρα. Για την αμοιβαιότητα. Εάν η Κίνα μπορεί να, να καταφέρει να αναλάβει την οικοδόμηση, την κατασκευή κομματιού αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Βαρσοβία και Βερολίνου, θα πρέπει και οι δικέ μα εταιρείε να μπορούν να κάνουν το ίδιο στου κινέζικου αυτοκινητοδρόμου, στου εξοπλισμού, στου σιδηροδρόμου. Ξέρετε ότι σήμερα αυτό είναι απολύτω αδύνατο. Οι αγορέ αυτέ είναι 100% κλειστέ στου Ευρωπαίου. Δεν στοχεύω την Κίνα ειδικώ αλλά εάν η καναδέζικη εταιρεία, η Bombardier, μπορεί στη Γαλλία να αναλάβει την κατασκευή ε, σειρμών, μάλλον γραμμών του μετρό και ε, αλλού, θα πρέπει και εμείς να μπορούμε να συμμετάσχουμε σε ανάλογους διαγωνισμούς στον Καναδά. Αυτό δεν είναι σήμερα δυνατό και αυτό δεν ονομάζεται αμοιβαιότητα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποδεχτεί κανείς τοικά αυτή την πραγματικότητα. Εμείς ως Ευρώπη είμαστε μια μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη. Παραμένουμε η πρώτη εμπορική δύναμη. Θα πρέπει λοιπόν την διαπραγματευτική μας πυγμή, να, η σχήμα, να την εκμεταλλευτούμε. Οι κινέζικες εξαγωγές προς την Ευρώπη είναι 280 δις ευρώ. Αντίστροφο είναι 150 οι ευρωπαϊκές εξαγωγέ προ την Κίνα. Δείτε τι διαφορά υπάρχει. Θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με τους Κινέζους και να του πούμε ε, και να το πετύχουμε και με αρκετή επιτυχία, διότι η κινέζικη αγορά με τις συνεχείς γαλλικές προσπάθειες ανοίγει λίγο-λίγο. Πολύ λίγο, με χαραμάδες μόνο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να ανοίξει αυτή η πόρτα. Δεν πρέπει να μας σταματήσει ούτε ο φόβος των αντιπίνων. Εάν δεν μπορέσουμε να κερδίσουμε ένα δημόσιο διαγωνισμό στην Κίνα, δεν θα πρέπει να δεχτούμε οι Κινέζοι να μπορούν να πάρουν μια δημόσια προμήθεια στην Ευρώπη. Δεν είναι περίπλοκο, είναι αρκετά απλό και θα είναι πολύ πιο δαπανηρό, θα είναι πολύ μάλλον λιγότερο δαπανηρό για τους φορολογουμένους μας να έχουμε εισαγωγή της ενεργείας. Διότι καλό είναι να προστατεύουμε τους καταναλωτές, αλλά θα πρέπει κάτι να κάνουμε και για τους παραγωγούς. Άρα, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι δικέ μα δημόσιες προμήθειε είναι πολύ πιο ανοιχτέ από ό,τι συμβαίνει με του ανταγωνιστέ μα. Όλα τα δεδομένα το αποδεικνύουν αυτό. Εμεί ω Ευρωπαίοι έχουμε πολύ λιγότερε δυνατότητε ε, να ανατρέξουμε στο ε, αμυντικό πλωστάσιο του ΠΟΕ από ότι οι βασικοί μα ανταγωνιστέ. Πολύ δυνατό, λιγότερε δυνατότητε ε, μέτρων πολύ λιγότερε δυνατότητε να τρέξουμε σε μέτρα anti-dumping ή κατά των επιδοτήσεων εφόσον χρειαστεί. Οι περισσότερε από τι εταιρείε, από τι μεγάλε αναδυόμενε οικονομίε, επιδοτούνται υπέρ των δέων με μεγάλο ποσοστό τίτλων και μας επιβάλλεται αθέμετος ανταγωνισμός, ο οποίος πλήττει και καταστρέφει ολόκληρα τμήματα της δικής μας βιομηχανικής παραγωγής. Για πόσο καιρό λοιπόν θα αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα κατάματα και να αντιδράσουμε. Το κείμενο που μας υποβάλλεται, κατά την άποψή μου, και σωστό προσανατολισμό έχει και σωστή έμπνευση. Η αμοιβαιότητα είναι η πρώτη κύρια αρχή που θα πρέπει να υπερισχύσει. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσω στο δυνατόν συντομότερη εξέταση του φακέλου διότι πραγματικά έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα ταχύτητας στις ε, ευρωπαϊκές χώρες. Η ο προστατευτισμός, είτε τον ονομάσουμε ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκό νόμο της διάσωσης ή όπως αλλιώς θέλουμε, ε, ή μάλλον by European ή ό,τι μάλλον μας αρέσει ε, θα πρέπει να λειτουργήσει. Ιδάλλως εμείς θα χάσουμε πρώτοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Λάγκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Επιτροπή αυτή έχουμε κάποια κοινά στοιχεία, αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά με τον κύριο Φελνερ που πρέπει να την τονίσω. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η απόφαση για μια δημοσία σύμβαση πρέπει να διαπέτει από την τιμή. Όχι, θέλουμε ποιότητα και όχι κοινωνικό ή dumping, μισθολογικό dumping. Κύριε Φέλνερ, και εσείς ε, ψηφίσατε μια έκθεση για την βιομηχανική πολιτική και είπαμε ότι στις δημόσιες συμβάσεις ε, θέλουμε να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια βιομηχανικής πολιτικής και να φέρουμε δύο κριτήρια. Θέλουμε την ενίσχυση της κοινωνία αφενός και αφετέρου θέλουμε να προωθήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα δύο κριτήρια δεν ε, επιτρέπουν να επιλέξουμε την πιο φθηνή προσφορά από όπου και αν προέρχεται, από την Κίνα ή αλλού. Όχι. Θέλουμε τα δημόσια χρήματα να χρησιμεύσουν για να ενισχύσουν τη δημιουργία θέσεων εργασία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για να γίνονται σεβαστά συγκεκριμένα πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αυτά τα πρότυπα, αυτά τα κανόνες να είναι καθορισμένα. αν ε, υπάρχει προσφορά και από άλλες χώρες ε, σε δημόσια συμβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτοί που υποβάλλουν τι προσφορέ θα πρέπει να σεβαστούν συγκεκριμένου κανόνε. Και αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα για να ξέρουν όλοι με τι έχουν να κάνουν. Δεν θέλουμε να συμβεί τι γίνεται σε άλλες χώρες που πολλές φορές δεν είναι γνωστά τα κριτήρια που διάβουν τις δημοσίες συμβάσεις. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια που θα ισχύουν όταν ανοίγουν οι δικές μας δημοσίες συμβάσεις και όταν ανατίθεται. Εμείς θέλουμε ποιότητα και σεβασμό συγκεκρισμένων ε, κανόνων και προτύπων και θέλουμε οι επιχειρήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου να ξέρουν ε, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να σεβαστούν. Κύριε Χέλμουντ, υπάρχουν παραδείγματα όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ε, προσφέρει υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα σε σχέση με το τι υπάρχει σε άλλες χώρες. το χάρη σε μια περίπτωση στο Καζακτα... Καζακστάν σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων, εκεί προσφερόνταν καλύτερες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν, αν ε, λάβουμε υπόψη τα κριτήρια της ποιότητας, πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτούμε και την εφαρμογή τους και πρέπει και να βρούμε και μηχανισμούς για την εκτελεσή τους. Εγώ δεν ξέρω αν ε, αυτό θα ε, εγκριθεί τελικά έτσι όπως έχει την νομοθετική πρόταση σήμερα. Μπορεί να υπάρξουν καλύτερες προτάσεις, αλλά δεν θα ήθελα ούτε και να βιαστούμε. Όπως ε, συμβαίνει και στην κίνηση, αυτό που μετράει δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ασφάλεια. Και καλή οργά παρά ποτέ. Δηλαδή, να προχωρήσουμε, αλλά να συζητήσουμε εις βάθος. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο σήμερα. Παρακαλώ, Φρανκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, συμφωνώ με όσα υπόθηκαν και είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε νομίζω ότι το να λέμε περισσότερα και να έχουμε περισσότερα κριτήρια είναι καλύτερο από το λιγότερο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα ρύθμιτο αριθμό χωρών που σήμερα δεν κάνουν καμία προσπάθεια για την αμοιβαιότητα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναφερθώ στην τελευταία περίπτωση που είχαμε προσφορά για το μετρό του Λονδίνου και είδαμε και την στάση της Ιαπωνίας. Επικεντρωθήκαμε αυτοκίνητο αυτοκινητομηχανία, αλλά υπάρχουν μια σειρά τομένων που βλέπουμε ότι η έννοια της αμοιβαιότητας δεν γίνεται σεβαστή. Όμω αυτό πηγαίνει πέρα και από τι δημόσιε συμβάσει. Στο Στρασβούργο την περσμένη εβδομάδα συζητήσαμε το dumping ε, στην περίπτωση τη Κίνα για τα φωτοβολταϊκά και ε, στη συνέχεια είχαμε και την υπόθεση της Ιλκόνης και τους γερμανούς παραγωγούς. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε σήμερα πράγματι να παίξουμε στους κανόνες της παγκόσμια αγοράς, μου φαίνεται καλό μεν, αλλά θα πρέπει όλοι να παίζουν με τους ίδιους κανόνες, όλες οι χώρες. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν ε, μπορούμε απλώς να δρούμε προληπτικά. Αν θέλουμε να γίνει σεβαστή η Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρχει μια Ευρώπη που να δρά και να προστατεύει. Και πιστεύω το να λάβουμε υπόψη μόνο τους καταναλωτής εν τέλει ε, δεν σημαίνει ότι τελικά τον προστατεύουμε να έχουμε χαμηλή τιμή αλλά υπάρχει μία σειρά ε, κανόνων ε, περιβαλλοντικών, μισθολογικών, εργασιακών που θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί για να προστατεύεται τελικά και ο καταναλωτής. Ευχαριστώ. Πίτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσω, αλλά θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό θέμα. Και ε, δεν πρέπει να συμβαστούμε με τους εθνικούς κανόνες, πρέπει να υιοθετήσουμε τους κανόνες του ΠΟΕ και να τους συμπληρώσουμε, να τους βελτιώσουμε με ε, διμερείς ε, συμφωνίες. Ο συνάδελφος μας είπε ότι επειδή είναι ο εισηγητής ε, για την ε, ε, σχέση με τον Καναδά, ελπίζω ότι το θέμα θα λυθεί με τον Καναδά. Αυτή είναι και η σωστή κατεύθυνση. Εγώ θέλω να επισημάνω και Κάτι άλλο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κοινή αγορά ε, δεν λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, κυρίως ε, για τις ε, μικρές συμβάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση, κυρίως ε, λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε τώρα, όπου διερχόμαστε κρίση με υψηλή ανεργία. Τώρα θέλουμε να επιταχύνουμε τις ε, συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με άλλες χώρες. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να δούμε τα του οίκου μας. Να βρούμε τους κανόνες που θα μας βοηθήσουν ε, να έχουμε ε, περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη να βγούμε από το αντιέξοδο. Ευχαριστούμε πολύ Πίτα και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και όλους ε, όσοι εξέφρασαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις επί του θέματος. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για μας, γιατί και εμείς επιθυμούμε να αντιδράσουμε σε κάποια από τα θέματα που ελέγχθησαν ε, σήμερα. Θα είμαι σύντομος, ε, θα ήθελα όμως να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι τι θα γίνει με τα άρθρα 58-59 που δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν. Προφανώς και πρέπει να είμαστε συνεπείς. Εφόσον προτείνουμε τέτοιου είδου εργαλεία, ε, ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί η πρόταση Κομισιόν. Ε, υπάρχει η οδηγία περί κοινοφελών οργανισμών. Ελπίζουμε ότι αυτό το θέμα θα περάσει. Και αργότερα ίσως αντιμετωπίσουμε κάποιες άλλες καταστάσεις. Ας τα αφήσουμε τώρα προς το παρόν. Ο κύριος Κάζακ έθιξε το ερώτημα το κατά πόσον είναι αντιφατικό να υπάρχει το 6 και το 8 ή το 10. Κοιτάξτε, εφόσον διαπραγματευόμεθα με τη Βραζιλία ή άλλες χώρες για να ανοίξουν την αγορά τους, παράλληλα, εφόσον υπάρχει ένας φορέας ε, που ζητάει τον, ε, κάποιον αποκλεισμό μιας ε, ε, συμφωνίας, ενός διαγωνισμού, είτε μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη μόχλευση ή να πει ότι αυτό ε, διαταράσει τις διαπραγματεύσεις. Μπορεί κανείς να το δει και από τις δύο απόψεις. Εμείς καταλήξαμε στο ότι στον κανονισμό υπάρχει προθεσμία. Εφόσον έχουμε λάβει απόφαση σε κοινοτικό επίπεδο, τότε ε, πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία. Θα μπορούσαμε να εξαιρέσουμε φορείς ευθύς εξ αρχής, αλλά δεν το κάναμε αυτό, γιατί θέλαμε να δώσουμε το μήνυμα στους εταίρους ότι είμαστε σοβαροί όσον αφορά το θέμα αυτό. Κατόπιν υπάρχει ένα περισσότερο φιλοσοφικής φύσης ερώτημα του κ. Ζαντό και άλλων, δηλαδή κατά πόσο είναι καλή ιδέα να υπάρχει αυτό το στοιχείο της βιομηχανικής πολιτικής στην πολιτική μας για ε, δημόσιες ε, προμήθειες συμβάσεις. Κοιτάξτε, η βιομηχανική πολιτική είναι αυτή που είναι, αλλά η πολιτική δημόσια συμβάσεων, εφόσον οδηγεί σε αυτό που είδαμε σε ορισμένε ε, χώρες ε, και εφόσον υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στόχοι που δεχόμαστε, ε, να υπάρχει ένας κανόνας όπου να είναι δεσμευτικό να αγοράζει κανείς επιτόπου τα υλικά, αυτό σημαίνει το τέλος του ελεύθερου εμπορίου. Ε, στον ΠΟ για πάρα πολλά χρόνια υπήρχαν κανόνες οι οποίες εξαιρούσαν αυτές τις πολιτικές ε, τοπικού περιεχομένου γιατί αν αρχίσει κανείς να λέει στους πολίτες του αγοράστε τα τοπικά προϊόντα ε, αυτό είναι αρνητικό κυρίως αν το πει στην Αμερική γιατί αν το κάνουν όλοι αυτό νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην εμπορική πολιτική. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κοιτάμε την αξία του χρήματος αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι κανονικά το επιχείρημα της αξίας του χρήματος ε, είναι σαφές. Ε, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο που δεν αναφέρθηκε και σε αντίδραση με αυτά που είπαν ο Κρίστοφ Βεάνερ και άλλοι. Τα μηνύματα που παίρνουμε τώρα από άλλους εταίρους είτε στη Γενέβη όπου ε, όλο και περισσότερες χώρες ζητούν υποβάλλουν διεκδικήσεις, οι άνθρωποι, ε, μάλλον το μήνυμα ότι είμαστε σοβαροί για το θέμα αυτό, κατά πόσο μπορούμε να ενθαρρύνουμε και άλλους να είναι πιο ανοιχτοί, αυτό το μήνυμα ήδη περνάει. Κατόπιν ετέθη ένα ερώτημα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες ή συγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης αντικτύπου. Εγώ δεν λέω ότι ότι αυτό σημαίνει υποστήριξη όλων των ε, στοιχείων. Από τις, ε, έχετε δίκηση στην εικόνα, η οποία είναι κάπως μεικτή, δηλαδή δεν έχουν αντιδράσει όλοι θετικά, αλλά σε γενικές γραμμές ε, πιστεύουμε ότι μας στηρίζουν. Η μελέτη αντικτύπων έχει το πρόβλημα του να ποσοτικοποιήσει τα θέματα, διότι δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα που να ε, συλλέγονται συστηματικά, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για ξένους μετέχοντες. Εμείς ε, έχουμε ε, συγκεκριμένα μοντέλα, αλλά δεν συμφωνούν όλοι επ' αυτών και ελπίζω έτσι απαντάτε το ερώτημα ότι δεν είναι τα στοιχεία 100% ποσοτικοποιημένα. Αν δει κανεί τι εξελίξει ε, τη ε, πρακτική στου δημόσιου διαγωνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, θα διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή η ανταγωνιστικότητα ε, της τοπικής βιομηχανίας αντιμετωπίζει περισσότερους περιορισμούς. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί με συγκεκριμένα παραδείγματα, μερικοί ε, υψώνουν δάχτυλο, αλλά εδώ υπάρχει θέμα και επίσης όσον αφορά την ελεύθερη ε, διακίνηση των ε, προϊόντων. Αυτό είναι ένα θέμα που προσπαθήσαμε να το λύσουμε ε, όπου υπάρχει ο κανόνας του 50% ξένο υλικό, αλλοδαπό υλικό, αλλά υπάρχει και ο κανόνας της προέλευσης που ισχύει στις και εξαγωγες γιατί κάποιος ε, πρέπει να εξετάζει την προέλευση στην ε, οικονομία που έχουμε σήμερα, αυτό είναι όλο και πιο δύσκολο. Κατόπιν, θα ήθελα να τοποθετηθώ στο ερώτημα σχετικά με την ανάπτυξη. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, ξερούνται από αυτές τις προτάσεις. Αν μπορούν να υποβάλουν προσφορά, αυτές μπορούν. Άρα δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Ίσως ε, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός αλλά σε ανάμεσα σε πολύ ανταγωνιστικές ε, αναδυόμενες οικονομίες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Κοιτάξτε, ε, δυστυχώς πολλές φορές υπάρχει αδιαφάνεια. Δηλαδή δεν είναι αλήθεια ε, με το να διαφυλάσει κανείς ε, ένα διαγωνισμό ε, στους τοπικούς μετέχοντες ότι με αυτόν τον τρόπο ε, διαφυλάσσει κανείς καλύτερα την αξία του χρήματος. Δεν είναι έτσι, γιατί ε, έτσι διευκολύνεται η διαφθορά και άλλες αρνητικές πρακτικές. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι δεν πρέπει να το προβάλλουμε ιδιαίτερα αυτό το επιχείρημα. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι προβάλλουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη. Νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφό μου να μιλήσει λιγάκι για, το, ε, για την κυβερνητική συμφωνία περί προμηθειών ε, και για την προστασία της κοινή αγοράς. Κοιτάξτε, μερικοί λέτε ότι η εναλλακτική λύση να μην κάνει κανεί τίποτα. Αλλά αυτό δεν είναι εναλλακτική λύση, γιατί με τον τρόπο αυτό όλο και περισσότερε χώρε θα ενθαρρυνθούν να κάνουν αυτό που ήδη κάνουν ε, και να βάζουν περισσότερου όρου και περιορισμού. Ε, στην Ευρώπη, σε τελική ανάλυση, ε, θέλουμε να ενθαρρύνουμε να, το να υπάρχει ένα άνοιγμα, δείχνοντας βέβαια ότι ε, και εμείς ε, δεν είμαστε ανοιχτοί πάντα για όλους και για όλα. Να σχολιάσω κάτι που είπατε για την πολιτική εσωτερική αγορά για τα άρθρα 58 και 59. Όπως ξέρετε, σήμερα τα άρθρα αυτά τα περιλαμβάνονται μόνο για τον ε, τομέα των ε, δημοσίων αγαθών. Παίρνουμε χάρη για τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε ε, και το νερό. Δεν έχουμε αυτού τους κανόνες της προτάσει για μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων. Γιατί όπω εξήγησε ο κ. συνάδελφο, θέλουμε όλου τους κανόνες να του σέβονται οι προσφέροντες από το εξωτερικό. Κάποια στιγμή το Κοινοβούλιο ήθελε να επανεισάγει αυτά τα άρθρα για να υπάρχει κάποια συνέπεια στι συνάφειε διαπραγματεύσει. Όμω αυτό θα σημαίνει ότι θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο στι διαπραγματεύσει για τη μεταρρύθμιση. Όμω προ στιγμή πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί σε αυτό το μέσο και όχι στο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, για τις ε, δύο προσεγγίσεις που έχουμε σε αυτό το μέσο, δηλαδή για το άρθρο 6 και την πιο γενική προσέγγιση που έχουμε στα άρθρα 8 και 10, αποκεντρωμένη προσέγγιση, πιστεύουμε ότι αυτές οι δύο προσεγγίσεις θα πρέπει να μείνουν ε, από κοινού, ε, είναι συμπληρωματικές και πολύ στενά συνδεμένες μεταξύ τους, γιατί η διαδικασία που προτείνεται στα άρθρα 6 8 είναι οι καθημερινές συμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις εθνικές οντότητες ε, και αν αντιμετωπίζαμε ουσιαστικές αρνήσεις σε καθημερινή βάση σε σχέση με συγκεκριμένε χώρες, τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το μέσο του άρθρου 10 ως ένα πιο γενικό μέτρο, αλλά πιστεύουμε ότι το ένα μέτρο χρειάζεται το άλλο, προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη συμμετοχή των ξένων προσφερόντων. Επίσης έγινε αναφορά σε αυτό το καθεστώς, κυρίως το καθεστώς του άρθρου 6 θα αυξήσει το κόστος ε, ε, για τα 60%. Ε, να υπενθυμίσω ότι στο σημερινό καθεστώς, το καθεστώς που έχουμε από το άρθρο 6, θα αποφασίσει η αρχή, η αρθέτους αρχή, αν θα αποκλείσει κάποιους προσφέρονται μπορεί και να καλέσει και προσφέροντες από χώρες όπως η Κίνα να συμμετάσχουν. Έτσι λοιπόν εξαρτάται από αυτούς και αν ε, για οποιοδήποτε λόγο ε, επιθυμούν να απορρίψουν κάποιο προσφέροντα τότε αυτό φυσικά θα επιφέρει διοικητικό άκθος αλλά δεν νομίζουμε ότι θα έχουμε αύξηση 60% του κόστους για την αναθέτουσα αρχή και άκουσα κάποια σύγχυση για τα δεδομένα. Θα πρέπει να το διορθώσουμε αυτό, εξηγώντα ότι σύμφωνα με τι δικέ μα εκτιμήσει, τα 5 εκατομμύρια ευρώ, το κατόφλι αυτό, σημαίνει ότι για όλε τι συμβάσει με αξία κάτω των 5 εκατομμύριων ευρώ θα έχουμε ανοιχτό διαγωνισμό και για του ξένου προσφέροντε. Αυτό σημαίνει 93% των συμβάσεων που είναι από δημόσια συμβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν το 93% θα είναι ανοιχτό και μόνο το 7% ε, μπορεί να τύχει προσωρινή άρνηση σε ό,τι αφορά την, ε, την αξία τη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ε, το 40% θα είναι ανοιχτό, αλλά το 60% μπορεί να εμπίπτει στο άρθρο 6 στην περίπτωση που ζητηθούν αρνήσει. Και να υπενθυμίσω και πάλι, και αυτό συνδέεται με τον κατακαιρματισμό τη εσωτερική αγορά. Τι κάνει αυτό το μέσο, τη αντίθεση με τη σημερινή κατάσταση, θέτει ομοιόμορφα κριτήρια σε κοινωνικό επίπεδο για τον χειρισμό των ξενών προσφερόντων. Έτσι λοιπόν, ε, πιστεύουμε ότι ευνοεί την ε, εσωτερική αγορά η πρόταση αυτή. Έχουμε το Φιλιτών 5 ε, εκατομμύρια ευρώ και δεν υπάρχει στην περιτούμαθησία αυτό. Επίση, λεπτομερό, μιλάει για με ποια ομοιόμορφα κριτήρια οι αναθέτουσε αρχε μπορεί να απορρίψουν τους αλλοδαπούς προσφέρονται και οπω είπα ουσιαστική αμοιβαιότητα η Κομισιόν θα έχει λόγο σε αυτό, θα αποφασίσει σε βάση ad hoc για το αν θα αποκλείσει ή όχι κάποιον και είναι αποδεκτή αυτή, αυτός ο αποκλεισμός θα γίνει ένα τεστ αμοιβαιότητας και έτσι θα έχουμε περαιτέρω εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση όπου έχουμε απόλυτο κατακριματισμό γιατί έχουμε αποκλίνουσες πρακτικές στα διάφορα Έχουμε κάποια που απορρίπτουν κάποιους αλλοδαπούς προσφέροντες και υπάρχουν κάποια όπου καλωσορίζουν ε, τους αλλοδαπούς ε, προσφέροντες. Έτσι λοιπόν έχουμε κατακριματισμό της εσωτερικής αγοράς. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, έχουμε σεβαστεί τους ε, εφιστάμενους ελληνικούς κανόνες και νομίζω ότι για τους λόγους αυτούς σημειώνουμε τον κατακαιρματισμό. Και κάτι για το, ε, για το GPA. Ε, φυσικά σεβόμαστε τις... Ε, ε, τη συμφωνία για τις κυβερνητικές προμήθειες Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με τη Συμφωνία Κυβερνητικών Προμηθειών, να υπενθυμίσω ότι έχουμε σεβαστεί τι διεθνεί μα υποχρεώσει και αυτέ που έχουμε συνάψει υπό τη GPA, υπό τη Συμφωνία αυτή Κυβερνητικών Προμηθειών και αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέτρα αγορά θα υπάρχουν και θα υπάρχει εγγυημένη πρόσβαση σε σχέση με τι αγορέ, που έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε σε μια αμοιβαία βάση και αυτό θα αντικατοπτρίζεται στην πρόταση, αν και οι αναθέτουσες αρχέ, ακόμη και αν έχουμε συμφωνήσει στον αποκλεισμό, μπορούν και πάλι να καλέσουν ε, προσφέροντό να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν ε, οι υποχρεώσεις ε, των εταίρων για την GPA, για τις συμφωνίες κυβερνητικών προμηθειών είναι πλήρως σεβαστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναντέλφους για τη σημερινή συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι η αγάπη προς τα ντόπια προϊόντα σταματά εκεί που αρχίζει η τσέπη. Ε, και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πολλές φορές ε, και στους δημόσιους διαγωνισμούς. Υπάρχει ένα θέμα ε, που αφορά περισσότερο την Επιτροπή κοινή Αγοράς. Πρέπει να διευκρινιστούν κάποια θέματα και έχοντας κατά νου την αμοιβαιότητα, ας πούμε το γερμανικό TGV μπαίνει και στη Γερμανία θα πρέπει λοιπόν και το γερμανικό ICE να μπαίνει και αυτό στη Γαλλία και στην Αγγλία. Αλλά εντάξει, αυτά είναι θέματα που αφορούν μια άλλη επιτροπή. Ε, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα. Ε, σήμερα κατέστη απόλυτα σαφές ε, ότι αν καταθέσουμε την έκθεσή μου πολύ γρήγορα και ψηφίσουμε, τότε θα ικανοποιηθούν αυτοί που θέλουν την ταχύτητα και αυτοί που θέλουν την αδράνεια και αυτοί θα είναι ευχαριστημένοι γιατί θα πάει το θέμα στο ε, Συμβούλιο και εκεί θα παραμείνει σε αδράνεια. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω να αφήσουμε κάποιες εβδομάδες έτσι ώστε να βρούμε κάποια λύση σε αυτό το θέμα και θα ήμουν ευγνώμων εάν ε, μπορούσαμε να παρακαλέσουμε την υπηρεσία του Κοινοβουλίου για μελέτες αντικτύπων να ξαναδεί αυτό το θέμα γιατί σήμερα σχολιάσαμε την Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών ε, θα προτείνω κάτι τέτοιο. Και προτείνω επίσης ε, σύντομα να σκεφτούμε ποιον θα καλέσουμε στην ακρόαση και θα χαιρόμουν εάν σε αυτήν την ακρόαση είχαμε χρόνο για να δούμε τις επιπτώσεις στην κοινή αγορά αλλά και στο άνοιγμα αγορών άλλων χωρών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Ε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ ως εισηγητής για τη σημερινή συζήτηση. Και θα ήθελα τώρα να πάμε στο επόμενο θέμα, το υπαριθμόν 20. Πάμε στην ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εμπορικές για το επόμενο για, τα μέσα εμπορικής ε, εργασίας. Άμυνας, με συγχωρείτε. Η Επιτροπή ίσως μπορεί να σχολιάσει την έκθεσή της ε, για να υπάρξει ε, μια σοβαρή συζήτηση. Θα ήταν σκόπιμο να είχαμε πάρει την έκθεση έγκαιρα, αυτό δηλαδή σημαίνει πριν από ένα χρόνο, και θα ήμουν ευτυχής ε, αν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούσαν να κάνουν σήμερα αυτήν την ε, έκθεση με PowerPoint. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να τελειώσουμε στις 6.30. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κύριους Βέλγιο και Μιούλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το θέμα λοιπόν αυτό στην ημερήσια διάταξη, τα μέσα εμπορικής άμενας, θα λέγαμε κατά πρώτον να δούμε τις ε, δυνατότητες προσφυγής τρίτων χωρών κατά των Ευρωπαίων των ενωσιακών εξαγωγών. Δηλαδή, όχι να δούμε πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μέσα εμπορική άμενα, αλλά πώ θα χρησιμοποιούν αυτά οι τρίτε χώρε και μάλιστα κατά των ε, εξαγωγέων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν κατά πόσον υπάρχουν έρευνες σε σχέση με αυτές τις εξαγωγές ή και μέτρα αυτά καθεαυτά. Η και μετρα αυτα αυτα προσφυγών και η μελέτη τους είναι μέρος της όλης μας δουλειάς για τη μελέτη της αγοράς και προκειμένου να παραμένουν οι αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοιχτές για τους εξαγωγείς μας. Εξάγουμε, διεξάγουμε monitoring, παρακολούθηση για να ενισχύσουμε τους εξαγωγείς μας και αυτό που θέλουμε να σα παρουσιάσουμε είναι μια κατάσταση των πραγμάτων όλη αυτή τη προσπάθεια παρακολούθηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει ετοιμάσει σχετική έκθεση, την ένατη κατά σειρά για την παρακολούθηση αυτή και η οποία απεστάλλει στο θεσμικό σα όργανο εγκαίρω. Πολύ σύντομα να πω ότι αυτό που θέλουμε να ε, καλύψουμε κατά πρώτον ε, είναι οι τάσει, θα δούμε κάποιου αριθμού, μετά θα δούμε τα βασικά προβλήματα, θα δούμε τα κύρια επιτεύγματά μας, τι έχουμε πετύχει σε αυτόν τον τομέα και τέλος θα δείξαμε κάποια συμπεράσματα. Κάποιες πρώτες τάσεις όταν ε, η αμυντική δράση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξαγωγών της μιας τρίτης χώρας ε, λαμβάνει χώρα, μας οδηγεί στην πρώτη σειρά αριθμών. Βλέπουμε εδώ το συνολικό αριθμό αμυντικών μέτρων κατά της Ένωσης και βλέπετε τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός ότι έχει παραμείνει σταθερός. Το 2009 είχαμε 138 περιπτώσεις, 123, το 2010 μια μικρή μείωση και το 2011 μια μικρή αύξηση. Περίπου όμως ένας ε, παρόμοιος συνολικός αριθμός. Εάν δούμε τώρα τις έρευνες που εκινήθηκαν κατά των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε μια παρόμοια τάση. Εάν δείτε στη δεξιά πλευρά του γραφήματος, 45 έρευνες εξήχθησαν το 2009, μειώθηκαν σε 40 το 2010 και ακόμη περισσότερο σε 33 το 2011. Μια περιορισμένη λοιπόν μείωση, αλλά η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς είναι ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει και όλα αυτά ε, φύλλονται στην δράση μας για τις ε, εγγύσεις, όχι τις διμερείς εγγύσεις, τις οποίες έχουμε συζητήσει διεξοδικώς ε, στο Κοινοβούλιο, αλλά δραστηριότητα διαφύλαξης μέσω των κλασικών μέτρων εγγύσεων τα μέτρα αυτά εξασκούνται όταν ε, μια χώρα αποφασίσει να διεξαγάγει έρευνα ή να ε, λάβει μέτρα για εξαγωγές από οποιαδήποτε πηγή. Εάν υπάρχει λοιπόν έρευνα εγγύησης, ε, το αποτέλεσμα που προκύπτει αφορά όλες τις εισαγωγές, είτε είναι από τις ΗΠΑ, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από την Ινδονησία ή οπουδήποτε αλλού με διαφορά, με, σε αντιδιαστολή με το ε, dumping και το CBD που είναι, ε, συγκεκριμένο, αφορούν συγκεκριμένες πηγές εισαγωγών. Βεβαίω πληττόμαστε γενικώ από τι εγγύησει. Ο όγκο εξαγωγών μα, δηλαδή, στη συγκεκριμένη χώρα που μπορεί να διεξάγει μια έρευνα ή λαμβάνει σχετικά μέτρα, μειώνεται. Στην Ινδία, λόγω χάρη, το 2009 είχαμε 10 έρευνε ε, εγγύησεων χωρίς να ληφθούν στη συνέχεια μέτρα, αλλά έτσι μειώθηκαν ε, ε, οι αριθμοί. Και γι' αυτό είχαμε 45 έρευνες το 2009. Ας δούμε τώρα τι υποκρύπτουν οι αριθμοί. Διότι οι αριθμοί είναι στοιχεία γυμνά, για να το πω έτσι. Τα προβλήματα που ε, υποκρύπτουν όμως, που υπόκεινται, είναι τα εξής στις τρίτες χώρες και στη δράση που αναλαμβάνουν στον τομέα αυτό, βλέπουμε ότι οι κανόνες του ΠΟΕ δεν γίνονται πάντοτε σεβαστοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εξασκεί αμυντικά μέτρα. Μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, αλλά τίποτα δεν μπορεί να κάνει για αυτά που λαμβάνουν τρίτε χώρε. Αρκεί βεβαίω να είναι νόμιμη η εξάσκησή του βάσει των διεθνών κανόνων όπω γνωριστεί στα πλαίσια του ΠΟΕ σε άλλε διεθνεί συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ανακύπτουν διάφορα προβλήματα. Το πρώτο είναι η ακατάλληλη χρήση των μέτρων. Αν σταθώ εδώ σε δύο επιμέρους παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα η, τα αντίπεινα. Ε, στο παρελθόν είδαμε περιπτώσεις αμυντικής προστασίας που ήταν ε, μια κλασική περίπτωση αντιπίνων. Αυτό ακολουθεί την εξή ε, διαδικασία συνήθω. Ανοίγει μια αμυντική υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόμοια υπόθεση ανοίγει μετά από λίγο στην τρίτη χώρα, κατά των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, μόλι ε, εντοπιστεί μια τέτοια υπόθεση, δεν μπορεί να γίνει κάτι, όμω ε, έχουν προκύψει πολλέ ε, συμπτώσει, οι οποίε είναι αρκετά παράξενες. Επέβαλε μέτρα κατά της εισαγωγής συγκεκριμένου τύπου αλεύρων από τρίτες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέσως έλαβε ανάλογα μέτρα και η τρίτη χώρα. Ε, για τα ανάλογα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κάτι ανάλογο έγινε και στην περίπτωση των σαρωτών, των σκάνερ που εισάγονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την τρίτη χώρα μετά άνοιξε επίσης έρευνα για, τους, για τα σκάνερ, τους σαρωτές που εισάγονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Ε, ξεκίνησε έρευνα και επέβαλε μέτρα για τις αντζούγες, για το γάβρο από συγκεκριμένες χώρες και μετά από λίγο η τρίτη χώρα μπόρεσε να ε, ανέλαβε παρόμοια μέτρα για το ίδιο προϊόν ε, όταν εισαγόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθούμε πολύ στενά τέτοιες περιπτώσεις. Κατά τη διεξαγωγή τη έρευνα παρεμβαίνουμε, συντονίζουμε την ενδιαφερόμενη, τον ενδιαφερόμενο βιομηχανικό κλάδο και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με τις χώρες που μπορεί να πλήττονται από αυτή την ε, έρευνα. Τα παρακολουθούμε όλα στενά, προκειμένου οι κανόνες να γίνονται σεβαστοί. Εάν όμως η υπόθεση είναι σοβαρή, σε τέτοια περίπτωση μπορεί να προστρέξουμε και στον ΠΟΕ, στο ανάλογο πάνελ επίλυση διαφορών στη Γενέβη. Μια τέτοια περίπτωση θα εξεταστεί του χρόνου. Η χρήση τώρα των μέσων ε, εγγυήσεων είναι ένα ιδιαίτερο αμυντικό μέσο. Το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις τρίτες χώρες. Είναι πολύ ευκολότερο από, να χρησιμοποιηθεί από τη, τα μέτρα διότι είναι λιγότερα κατακριτήρια που χρειάζεται να ενεργοποιηθούν εδώ και μπορεί να ισχύει ταυτόχρονα για όλες τις εισαγωγές από όλες τις πηγές εκτός της τρίτης χώρας. Πολύ συχνά άλλωστε το πρόβλημα ε, που αφορά μια συγκεκριμένη έρευνα διερεύνησης εγγυήσεων έχει να κάνει με μία ή δύο το πολύ χώρες. Και ενώ αρχικό στόχο είναι ο μία ή δύο χώρε, τελικά το πρόβλημα δεν επεκτείνεται και αφορά και όλου του υπόλοιπου. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη διαφάνεια. Κάτι ε, που συστηματικά προκύπτει. Εάν ένας εξαγωγέας ε, είναι αντικείμενο έρευνας ε, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και η αρχή που είναι επιφροντισμένη με την έρευνα αποφασίζει πρέπει να αναλυθούν μέτρα, τότε ο εξαγωγέας δεν θα ξέρει ακριβώς πώς το περιθώριο του ντάμπινγκ έχει υπολογιστεί από την ερευνητική αρχή. Θα το ξέρουν δεν μπορούν να ξέρουν μάλλον οι εξαγωγείς ή οι συνηγοροί του γιατί το δεκαδικό ψηφίο μετά την υποβιαστολή είναι ο τάδε ή ο τάδε αριθμός. Υπάρχουν χώρες βέβαια που είναι αδιαφανείς τις διαδικασίες αυτές και δεν είναι και τόσο ανεπτυγμένες. Κανείς δεν μπορεί λοιπόν από τους εξαγωγείς να γνωρίζει πώς το περιθώριο του ντάμπινγκ έχει υπολογιστεί και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις ερευνητικέ αρχές των τρίτων χωρών να εφαρμόσουν πρότυπα. Πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν μια κάποια διαφάνεια. Τελευταίο πρόβλημα που έχω εντοπίσει ε, για την παρουσίαση αυτή είναι η εντυνόμενη περιπλοκότητα. Στο πρόσφατο παρελθόν είδαμε ότι η αξία των εξαγωγών που έχουν επηρεαστεί από τέτοιε είναι, περιπτώσεις είναι αρκετά σημαντική. Φτάνουν το επίπεδο των δισεκατομμυρίων. Και στην Ένωση υπάρχουν βέβαια αναλλαγές υποθέσεις που επηρεάζουν σημαντικό όγκο σημαντικό όγκο συναλλαγών, εμπορικών συναλλαγών. Απλώ οι υποθέσει γίνονται όλο και πιο περίπλοκε λόγω των ζητημάτων που εξετάζονται. Ιδίω για υποθέσεις που έχουν να κάνουν και με τη χρήση των εργαλείων επιδοτήσεων. Διότι εάν είναι εκτεθειμένη προς κάτι τέτοιο η Ένωση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συντονιστούν οι εξαγωγείς των οποίων βρίσκονται στο στόχαστρο οι συγκεκριμένε εξαγωγές αλλά και το συγκεκριμένο σύστημα επιδότησης. Είτε αυτές που έχουν εγκριθεί από την ίδια την Ένωση είτε αυτές που έχουν εγκριθεί από τους κατοικούς νόμους επιδοτήσεων, από τα κάτι μέλη δηλαδή. Χρειάζεται ένας μεγάλος βαθμός συντονισμού. Και βεβαίως η ζωή μας γίνεται πιο περίπλοκη. Μίλησα τώρα για προβλήματα, αλλά ας πούμε και τα επιτεύγματα. Πέρυσι είχαμε μια επικοδομητική χρονιά με πολλά θετικά αποτελέσματα. Ένα ήταν η περίπτωση του μεδενισμού. Ξέρετε ότι για, την, ε, για τον απολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ εξασκούν το μέτρο αυτό οι Ηνωμένε Πολιτείε και πολλά μέτρη του, μέλη του ΠΟΕ είχαν αντιταχθεί στην πρακτική του zeroing αυτού, του μηδενισμού των ΗΠΑ, τελικά όλα αυτά είχαν αίσιο πέρας. Αλλά υπήρχαν και συγκεκριμένε υποθέσεις. Έκλεισαν συγκεκριμένε υποθέσεις. Όπως ε, μία που ε, αφορούσε την Ουκρανία και μέτρα dumping για πετρελαϊκά προϊόντα. 500.000 ευρώ εξαγωγές, 500 εκατομμυρίων ευρώ αξίας οι εξαγωγές. επηρεάζονταν κυρίως η Πολωνία. Αλλά με συντονισμό των πολωνικών και λιθουανικών αρχών Ε, και χάρη στις σχέσεις με την Ουκρανία, οι εξαγωγές προς τη χώρα αυτή τελικά σώθηκαν. Επίσης υπήρχε μια υπόθεση που αφορούσε ψυγεία, μια άλλη που αφορούσε κρασί, τον Ίνο, υπόθεση που έκλεισε τον Οκτώβριο, με αφορούσε την Βραζίλια και βεβαίως προηγουμένως υπήρξε ενδονοσιακός συντονισμός Προστατεύσαμε έτσι τι εξαγωγέ μα, αλλά είχαμε και πολύ καλό συντονισμό με άλλε τρίτε χώρε που αφορούσε συγκεκριμένη έρευνα, η έρευνα τη Βραζιλία αυτή, τι ΗΠΑ, την Αζηλανδία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νότια Αφρική. Μεταξύ άλλων. Υπάρχουν και άλλα δύο παραδείγματα. Αυτά είναι επιτεύγματα που πετύχαμε, δεν είναι μόνο λοιπόν ζωφερή εικόνα, κάποιε φορέ είναι και φωτεινότερη. Και εδώ στην τελευταία διαφάνεια Έχετε ορισμένα συμπεράσματα, συμπεράσματα τα οποία συνέταξα. Είναι εντατικέ οι δράσει που αναλαμβάνουν στον τομέα αυτό οι τρίτε χώρε. Αυτό που χρειάζεται είναι βεβαίω συντονισμένε προσπάθειε στον όλο τομέα. Κάναμε λόγο για την ε, περιπλοκότητα λόγω του οικονομικού όγκου, αλλά και μην, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τον ε, καθοριστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορεί να κινητοποιήσει τους ενδιαφερομένους και τους εμπλεκομένους για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους εξαγωγείς. Θα ήθελα να κλείσω εδώ λόγω και της ώρας που έχει περάσει πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και το ερώτημα που ε, θέλω να κάνω είναι μήπως επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο επί του θέματος. Αν ε, δεν ε, ισχύει αυτό, τότε θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παρατήρηση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την Ολομέλεια στο Στρασβούργο και εκεί ε, μιλήσαμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση anti-dumping. Νομίζω ότι πολλοί στη συζήτηση συμφώνησαν ότι θα χαιρόμασταν η Κομισιόν να μην εκμεταλλευτεί το μέγιστο χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεσή της ε, για εξέταση και ε, νομίζω ότι επειδή δεν θα είναι ο Επίτροπος παρόν ε, θα ήμουν ευγνώμων η Κομισιόν να εξετάσει αυτό το θέμα και η Γενική Διεύθυνση και εσείς ότι θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Θέλετε να πείτε κάτι. Αν δεν υπάρχουν... Ε, α, μισό λεπτό. Ο Γιάννικ. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου θα είναι σύντομη. Για τους οικολόγους, ένα σημαντικό θέμα που θα θέλαμε να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτό που αφορά την ε, αντιμετώπιση των, και την εξέλιξη των επιδοτήσεων. Το είδαμε και το θύμισε ο κύριος Κάσπαρη για το θέμα των ε, φωτοβολταϊκών από την Κίνα. Αυτό όμως που θέλουμε να μάθουμε είναι πώς εξετάζει το θέμα των επιδοτήσεων αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδίω των επιδοτήσεων που μπορεί να είναι αρνητικέ για το περιβάλλον. Το συζητήσαμε σε σχέση με την αλλήλεια αυτό. του Ε. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε αν έχει την πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει περιβαλλοντικά πρότυπα στα μέτρα αυτά προστασίας και αν πρόκειται να τα ενσωματώσει τα πρότυπα στα μέτρα προστασία. Υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη συζήτηση όταν μιλάμε για αντιμετώπιση των κλιματικών λαγών, λόγου χάρη ή για την διαφυγή του άνθρακα. Και λέμε πάντοτε ότι αν έχει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να προστατευτεί και από χώρε που προφανώς δεν επιβάλλουν παρόμοιες συμβάσεις TS στις επιχειρήσεις τους. Πόσο έχει λοιπόν προχωρήσει σχετικά η δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της συμπερίληψης περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων στην όλη εξέταση του θέματος των επιδοτήσεων και στο πώς ε, εξασκούνται οι επιδοτήσεις από τα κάτι μέλη. Δηλαδή, στην αντιμετώπιση των επιδοτήσεων. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό όμω, Πριν να φτάσω στις απαντήσεις, έχω και άλλη μια ερώτηση ως ε, μέλος. Υπάρχουν έρευνες στην Κομισιόν σχετικά με τις ε, επιπτώσεις ε, που έχουν περιπτώσεις ε, αντι-dumping, εξέταση αυτών των περιπτώσεων για τους απασχολούμενους στην Ευρώπη. Γιατί προβλέπεται στις αρχές του επόμενου έτους να ασχοληθούμε με την οδηγία αντι-dumping. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον για πολλούς από εμάς να γνωρίζουμε ποια είναι η εμπειρία με τις περιπτώσεις αντι-dumping και τι έχει υπάρξει συγκεκριμένα για τους απασχολούμενους και τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Ε, είναι εδώ και ένας άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μπέκερ που θέλει να παρέμβει για τις ερωτήσεις αυτές και να δούμε σε ποιο βαθμό θα απαντήσει. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την περιβαλλοντική και κοινωνική πτυχή της εμπορικής άμυνας. Η απάντηση σε αυτό ίσως να μην είναι ικανοποιητική κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όταν χρησιμοποιούμε τα παραδοσιακά μέσα εμπορικής άμυνας όπως είναι το anti-dumping ή το να μην χορηγούμε επιδοτήσεις, δεν υπάρχει διεθνής νομική βάση για να συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο στις δικές μας υποθέσεις. Λοιπόν, ε, δεν μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και να πούμε ότι εμείς ε, στην Ένωση έχουμε ένα επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ε, και αυτό είναι ακριβό. Και θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό στα αριθμητικά στοιχεία των Ευρωπαίων παραγωγών. Όμως αυτές οι δαπάνες δεν είναι απαραίτητες σε τρίτες χώρες που δεν έχουν τα ίδια πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας. Τώρα φυσικά υπάρχει ιδέα, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αυτό μέσω των διεθνών διαπραγματεύσεων. Αλλά προς στιγμή, ναι, έτσι όπω είναι τα κείμενα του ΠΟΕ και έτσι όπως είναι οι συμφωνίε, σε έναν υπολογισμό dumping δεν μπορεί να το λάβει υπόψη αυτό. Έτσι λοιπόν, την επόμενη ημέρα θα καταφερόταν κάποιο εναντίον μα στον ΠΟΕ, αν το προσπαθούσαμε και υπερβαλλοντικές ε, ε, σκέψεις. Η προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσε να συμπεριληφθεί αν είχαμε υπόθεση και καταλήγαμε στο συμπερασμά ότι έχουμε μια κατάσταση dumping ή χορήγησης επιδητήσεων και έχουμε ένα συμφέρον της Ένωσης, έτσι όπως το αποκαλούμε. Και ουσιαστικά έχουμε το ερώτημα, έχει νόημα να επιβάλλουμε τα μέτρα αυτά ή θα ήταν επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη τον περιβαλλοντικό σκέλος, αλλά ουσιαστικά αντίστροφα συμβαίνει. Και για να στραφώ στην ερώτηση του κ. Κασπαρή. Αφού έχουμε βάλει μέτρα, υπάρχει συνέχεια. Συστηματικά δεν προβαίνουμε σε follow-up, αλλά συνήθως επιβάλλουμε μέτρα για πέντε έτη και αυτά τα μέτρα μετά από πέντε έτη θα μπορούσαν να επιμηκυνθούν, να παραταθούν, αλλά γίνεται κάτι τέτοιο μόνο αν το ζητήσει η βιομηχανία, ο κλάδος που έχει κάνει την καταγγελία. Και αν υπάρχει μια τέτοια αίτηση, τότε έχει νόημα, θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία αναθεώρησης και σε αυτή την αναθεώρηση θα δούμε πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέτρα. Αυτό είναι το πιο πιθανό πιο πιθανή κατάσταση στο οποίο θα, στην οποία θα το εξετάζαμε. Πέραν αυτού, η γενική μας αρχή είναι ε, ότι αν υπάρχει ζήτηση, αναλαμβάνουμε δράση. Και καθώς συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνήθως χρειάζεται καταγγελία από τον αρμόδιο κλάδο, την αρμόδια μηχανία, θα πρέπει να έχει κάποιο κύρος και ουσιαστικά να καταγγείλει ότι έχει υποστεί ζημία και κατόπιν θα ανοίξουμε την υπόθεση αυτή και ακολουθούμε την ίδια κατάσταση. Αν μια Ευρωπαϊκή Βιομηχανία έρθει και μας πει μας ότι είναι αναπαρκή η προστασία, τότε θα αναθεωρήσουμε την υπόθεση. Αν έρθουν οι εξαγωγεί και μα πούνε είναι πολύ ψηλή δασμοί, ουσιαστικά αποκλειόμαστε από αυτή την αγορά και επίσης ε, αν υπάρχουν αποδείξεις θα προβούμε σε αναθεώρηση, αλλά γίνεται κατόπιν ετήσιο πάνω κάτω. Από την άλλη πλευρά δεν είμαστε τυφλοί στον διάμεσο. Έχουμε σχετικά καλή πρόσβαση στα ταστικά στοιχεία των εισαγωγών και έχουμε και μια ειδική στατιστική που δημιουργείται βάσει του βασικού μας κανονισμού, του άρθρου 14.6 όπου ε, τα τελωνία μας υποβάλλουν αναφορές σε σχέση με τους δασμούς που συλλέγονται για υποθέσεις αντι-dumping και μετά την, τις εισαγωγές μπορούμε να δούμε αν τα μέτρα ήταν αποτελεσματικά Δηλαδή βλέπουμε πώς εξελίσσεται ο όγκος αυτού του προϊόντος ε, αν έχουν δασμοί δεσμοί αντι-dumping. Μια άλλη δυνατότητα να δούμε τι γίνεται στην αγορά είναι Έχουμε την ε, παράκαμψη δηλαδή, μπορούμε να δούμε αν έχουμε τέτοια μοντέλα και στις στρατηγικές ε, εισαγωγής ε, βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, αν θα πρέπει να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση, αν τα μέτρα που επιβάλλουμε ε, τι κάνουν για την ευρωπαϊκή αγορά και την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Είχαμε και την πράσινη βιβλία του Επιτροπού Βάντελσον στο παρελθόν και μπορώ να σας πω ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες βασικά είπαν ότι δεν το θέλουν αυτό και σχεδόν χωρίς καμία διαφωνία. Και ο λόγος είναι απλός, γιατί τους κοστίζει πολύ, γιατί μπορεί κάποιος να αξιολογήσει την ε, ανάπτυξη της βιομηχανίας, αν υλοποιεί την ίδια έρευνα που έκανε αρχικά. Έτσι λοιπόν, αν έπρεπε να κάνεις άλλη μία έρευνα ζημία, σημαίνει ότι στέλνεις ερωτηματολόγια στους ευρωπαίους παραγωγούς, στους χρήστες, στους καταναλωτές, στους αγωγείς και υλοποιείς μία έρευνα και καταλήγεις στο ίδιο συμπέρασμα ή αλλάζει συμπεράσματα. Πέρα από το γεγονό ότι πιθανότητα δεν θα είχαμε του πόρου για κάτι τέτοιο. Και μία σαφής απάντηση από την Ευρωπαϊκή είναι ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο. Και πιστεύει ότι αρκεί οι εξαγωγή, οι ή οι άλλοι συμμετέχοντε στην αγορά που ενδιαφέρονται να παρουσιαστούν και να πούν συμβαίνει κάτι που είναι μη ικανοποιητικό. Και κάτι τελευταίο η ανησυχία ότι μπορεί να επιβάλλουμε πολύ ψηλού δεσμού. Δηλαδή, σε σύγκριση με το ΙΣΥΠΑ είναι πολύ χαμηλότεροι δεσμοί. Θα το ξέρετε αυτό. Αλλά σε αντίθεση με άλλε χώρε, εμεί έχουμε ένα επιπλέον εργαλείο υπολογισμού, τον κανόνα μικρότερου δασμού. Δηλαδή, όταν υπολογίζουμε ένα περιθώριο dumping, έχουμε και μια δεύτερη εξέταση αν χρειάζεται αυτό το πλήρες περιθώριο. Αν αυτό το πλήρες περιθώριο δεν χρειάζεται ε, για την άρση της μίας τότε επιβάλλουμε έναν χαμηλότερο δασμό. Δηλαδή, πράττοντά το αυτό συστηματικά και περισσότερο από το ίμιση των βασίζονται σε αυτόν τον υπολογισμό του χαμηλότερου δασμού, η πιθανότητα να ε, είναι υπερβολικά τα δικά μας μέτρα, τουλάχιστον ε, σε σχέση με άλλους χρήστες του συστήματος, είναι πιο περιορισμένη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο υπάρχουν. Όχι. Να σας πω ότι θα σας μοιράσουμε και την παρουσίαση PowerPoint τις επόμενες ώρες. Θα ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτηση. Αυτό θα συνεισφέρει στι ε, επόμενε συζητήσει που θα έχουμε το επόμενο έτος για τα μέσα εμπορική άμυνα. Θα οργανώσουμε και ένα εργαστήριο για το πλάσματα τη δημόσια διαβούλευση για το θέμα σε σχέση με την επόμενη συναντησίνητα στι 18 Δεκεμβρίου. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την έλευση σα εδώ σήμερα. Και να περάσω στα διάφορα. Σημείο 21. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις. Περνάμε στο σημείο 22. Προσέχει συνεδρίαση 17 και 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας σήμερα. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία. Πρόεδρος, ευχαριστώ και τους Και σας ε, εύχομαι να ε, ξεκινήσει ωραία χριστουγεννιάτικη περίοδος από την 1η Δεκεμβρίου.